So, guten Morgen, liebe und Kollegen. Καλημέρα, συνάδελφοι. Καλώ ήρθατε στην τελευταία συνεδρία πριν τι διακοπέ. Καλό είναι το ότι εμφανίστηκαν και μερικοί βουλευτέ. Σήμερα έχουμε βαρύ πρόγραμμα με την παρουσίαση της Πολωνικής Προεδρίας και καλωσορίζω τον κύριο Μάρεκ Σαβίτσκι, Υπουργό Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Πολωνίας, που έχει την Προεδρία. Και επειδή πέρα από την προστασία του περιβάλλοντος είμαστε αρμόδιοι και για τα τρόφιμα, υπάρχουν κάποια πράγματα να μας πει εδώ πέρα ο κύριος Υπουργός. Ο κύριος Υπουργός σπούδασε γεωπόνος, έκανε το διδακτορικό του επίσης στον ίδιο τομέα, ήταν γενικός γραμματέας στο Υπουργείο, αρμόδιο στο Υπουργείο Επικοινωνιών και είναι επίσης και ο ίδιος αγρότης. Δεν μιλάει μόνο για αυτά τα πράγματα. Και από το 1993 είναι βουλευτής στην Πολωνία και είναι επίσης πρόεδρος της Επιτροπής για την Προστασία του Καταναλωτή και τον Ανταγωνισμό και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος των Πολωνών Αγροτών. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Είχαμε την ευκαιρία και στη Βαρσοβία να τα πούμε και με ενδιαφέρον θα ακούσουμε τι σχεδιάζει η Πολωνική Προεδρία. Οπότε αναμένουμε την παρουσίασή σας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που μου δίνετε ευκαιρία να σας παρουσιάσω σήμερα τις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας για τη Γεωργία, την ανάπτυξη της Πέθρου και την Ελία. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τη δυνατότητα που μου δίνετε και πρώτα απ' όλα να ευχηθώ στους Γάλλους Ευρωβουλευτές για την εθνική τους εορτή και όπως είπε και ο Πρόεδρος, μια και είναι τελευταία ημέρα των, των συνεδριάσεων, καλές διακοπές. Ε, γι' αυτό δεν είναι και κανείς εδώ πέρα, τέλος πάντων είναι τόσο λίγοι. Κυρίες και κύριοι, η Πολωνία είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία η γεωργία εξακολουθεί να έχει τεράστια σημασία. Γι' αυτό και η Πολωνική Προεδρία έχει ως προτεραιότητες την ασφάλεια της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, την ενέργεια και την άμυνα. Και το θέμα των τροφίμων, η ασφάλεια τροφίμων βρίσκεται ε, στην πρώτη θέση των προτεραιοτήτων μας. Είδαμε τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες ε, τη τεράστια σημασία έχει για όλους μας η ασφάλεια των τροφίμων. Και όταν λέμε ασφάλεια των τροφίμων ε, μπορούμε να την εννοήσουμε με πολλούς και διάφορους τρόπους. Καταρχήν η ασφάλεια της ποιότητας, η ασφάλεια της ποσότητας, αλλά ταυτόχρονα και η ασφάλεια του ίδιου του παραγωγού των τροφίμων που πρέπει να προγραμματίσει, να προσχεδιάσει τις δραστηριότητές του σε ένα πιο μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Σε ό,τι αφορά τη γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου, η Πολωνική Προεδρία θα επικεντρωθεί κυρίως στη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής μετά το 2013. Και σημαντικό στο μέσα εδώ θα είναι η συζήτηση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα ήθελα να επισημάνω ιδιαίτερα το σημείο αυτό, γιατί πριν από 150 χρόνια η γεωργία ήταν ε, αυτάρκης τομέας από ενεργειακή άποψη. Σήμερα όμως ε, εξαιτίας και των προκλήσεων που έχουμε για την προστασία του κλίματος, ε, του περιβάλλοντος και των κλιματικών αλλαγών είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με το θέμα της ενεργειακής αυτάρκειας των ε, Γεωργών και πάλι και εκεί το θέμα της βιομάζας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποκτά ιδιαίτερη σημασία και γι' αυτό αποτελεί προτεραιότητα και για μας. Και μάλιστα στα τέλη της εβδομάδας στο Σόποτ ε, το Σάββατο θα έχουμε συνάντηση για να εξετάσουμε ακριβώς αυτό το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ευελπιστώ ότι στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο θα μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε κάποια συμπεράσματα για το θέμα αυτό. Επίσης, ε, θα ήθελα στα πλαίσια των προτεραιοτήτων να αναφερθώ και στην κοινή αλλιευτική πολιτική, γιατί και η κοινή γεωργική πολιτική και η κοινή αλλιευτική πολιτική πρόκειται να μεταρρυθμιστούν. Και το τελευταίο τριήμερο στις ε, επαφές και συνομιλίες που είχα με τους ε, ευρωβουλευτές διαπίστωσα ότι υπάρχει επιθυμία για ρηξικέλευθη και βαθιά μεταρρύθμιση και της κοινή ελευτικής πολιτικής αλλά και για την κοινή γεωρική πολιτική. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρέ ανησυχίε και φόβους. Γιατί ναι μεν στην αλληλευτική πολιτική έχουμε ένα μεταρρυθμιστικό κίνημα που επικρατεί, ενώ στην γεωργική πολιτική έχουμε περισσότερο ένα ρεαλιστικό κίνημα. Πάντω στην αλληλευτική πολιτική υπάρχει σημαντικό αίτημα για ρηξικέλευτη μεταρρύθμιση, ενώ στην γεωργική πολιτική υπάρχουν περισσότερε ανησυχίε. Τώρα για τα υπόλοιπα ζητήματα θα ασχοληθούμε με το θέμα της ταυτοποίησης των βοηδών Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα την ε, πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ηλεκτρονική ταυτοποίηση των βοηδών. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια πλούστευση του μηχανισμού και ευελπιστώ ότι το Κοινοβούλιο ε, θα υποστηρίξει ε, την πρόταση του Συμβουλίου, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξουν την πρόταση του Συμβουλίου για απλούστευση. Στο θέμα της ταυτοποίησης των βοηδών ε, θα πρέπει να μας οδηγήσει και στην ε, ανάγκη ε, να εξετάσουμε και την ταυτοποίηση των προβάτων, γιατί το κόστος αυτής της ταυτοποίησης δεν είναι ανάλογα με τις απειλές αλλά και με την αξία των συγκεκριμένων κοπαδιών. Άλλο σημαντικό θέμα για την Πολωνική Προεδρία είναι η ευζοία, η ευημερία των ζώων. Γι' αυτό και περιμένουμε τόσο Θηνόπορο μια πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευημερία των ζώων και ιδιαίτερα τη μεταφορά. Πιστεύουμε ότι όλα τα θέματα, όλες οι πτυχές για την ευημερία των ζώων αλλά και οι οικονομικές πτυχές θα συμπεριληφθούν στον προβληματισμό, θα γίνει μια σωστή στάθμιση και θα καταλήξουμε σε ισορροπημένες ρυθμίσεις και λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις ε, ανησυχίε μας και το μέλημα για την ευημερία των ζώων, αλλά θα ανταποκρίνονται και στις οικονομικές ε, και περιβαλλοντικές μας δυνατότητες και ανησυχίες. Θα πρέπει να τα συμφιλιώσουμε αυτά. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια και για τα φυτοϊγειονομικά ζητήματα. Οι φυτοϊγειονομικές διατάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησαν πριν από μία τριακονταετία και νομίζω ότι είναι και η ώρα να προβούμε σε μία αναθεώρηση αυτών των φυτογειονομικών διατάξεων που είναι πια παροχημένες γιατί και ως προς τις νόσους, επιζωτίες, παράσιτα και παθογόνους παράγοντες έχουμε πολλές εξελίξεις. Είναι λοιπόν αναγκαία σήμερα μια αλλαγή αυτών των φυτογειονομικών κανόνων. Επίσης θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε και να απλουστεύσουμε τις νομοθετικές διατάξεις ό,τι αφορά την εμπορία των σπόρων και του πολλαπλαστικού υλικού των φυτών. Χρειαζόμαστε εναρμονισμένη και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά με υψηλή ποιότητα σπόρων αλλά και πολλαπλασιαστικού υλικού των φυτών. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προστατεύσουμε και το περιβάλλον και να λάβουμε υπόψη την όλο και μεγαλύτερη παγκοσμιοποίηση και την ανάγκη εφαρμογή διεθνών προδιαγραφών. Και στου δύο αυτού τομείς η Πολωνική Προεδρία θα συνεργαστεί στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι προπαρασκευαστικές εργασίε για τι νομοθετικέ προτάσει. Άλλο σημαντικό θέμα που σίγουρα θα μας απασχολήσει και ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες είναι το θέμα των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών η Πολωνική Προεδρία προτίθεται να συνεχίσει τις εργασίες για το πολύ σημαντικό αυτό το θέμα ε, που απασχολεί την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ώστε να δημιουργήσουμε πρόσφορο έδαφος και να καταλήξουμε σε τριμερή διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί η συζήτηση για το πρόβλημα αυτό μέχρι στιγμής που έχει γίνει στην Ευρώπη κατά τη γνώμη μου δεν είναι πλήρης. Υπάρχουν πολλά κενά στη συζήτηση που έγινε. Το 2011 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε το έτος αυτό Διεθνές Έτος των Δασών. Στην Πολωνία το 30% της επικράτειας καλύπτεται από δάση. Από αυτή την άποψη η βιοπικιλότητα σε εμά, ε, χάρη στα δάση, είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Το θέμα των δασών λοιπόν είναι κατά τη γνώμη μας πολύ σημαντικό ε, για το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Γι' αυτό και θα ήθελα να πω δύο λόγια και για τα δάση. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την προστασία των δασών και την ενημέρωση για τα δάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι βέβαιος ότι το Συμβούλιο θα ενστερνιστεί τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα υιοθετήσει μια υποφελή θέση για το περιβάλλον. Τα δάση έχουν και κοινωνικό χαρακτήρα και συμβάλλουν στην ε, οικονομική ανάπτυξη και τη υπαίθρου. Γιατί είναι πραγματικά φύλακες ε, των... Ε, οι φύλακε τη της και της προστασία του περιβάλλοντο σε μεγάλο βαθμό στον κόσμο είναι οι γεωργοί και οι δασοκόμοι. Η καλή κατάσταση των δασών, η αηφορία των δασών στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό. Ε, σημαντική είναι και η ενημέρωση για τους δασικούς πόρους της Ευρώπης. Όλα αυτά τα θέματα απαιτούν ακόμη καλύτερη προετοιμασία και συντονισμό στα πλαίσια και της προσπάθειας καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών. η πρώτη της ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτυχε ευρεία υποστήριξη και από τα κοινωτικά θεσμικά όργανα αλλά και από την κοινή γνώμη και θα συνεχίσουμε τις εργασίες σε συνεργασία ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά τα δάση θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Πολωνική Προεδρία θα συνεχίσει την εξαιρετική προσπάθεια που ξεκίνησε η Ουγγρική Προεδρία. Έχουμε το σχέδιο ε, τα δάση της Ευρώπης και υπουργική ε, διάσκεψη με θέμα την προστασία των δασών. Τον Ιούνιο στο Όσλο οι Ευρωπαίοι Υπουργοί για τα, Αρμόδιοι για τα Δάση έλαβαν σημαντική απόφαση για την έναρξη διαπραγματεύσεων σε ό,τι αφορά μια υποχρεωτική συμφωνία για τα δάση στην Ευρώπη. Επίσης ε, καθόρισαν τους ε, ευρωπαϊκούς στόχους μέχρι το 2020 για τα δάση. Η πρώτη διαπραγματευτική σύνοδος ε, για ε, ένα υποχρεωτικό κανονισμό έχει προγραμματιστεί για το Νοέμβριο του 2011. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η, αυτή η υπουργική συνδιάσκεψη να ετοιμαστεί και να διοργανωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα υπάρχει και η Παγκόσμια Οργάνωση για το, το τροπικό ξύλο. Θα πρέπει να διεκπαιρεθούν οι διαπραγματεύσει για τη σύναψη, ε, για την κύρωση της σύμβασης ε, που ε, υπογράφηκε το 2006. Η Πολωνία πρόκειται να συνεργαστεί στα πλαίσια της Προεδρίας της με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα κράτη-μέλη. Θεωρούμε ότι μετά τη δημοσίευση της έκθεσης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται να εγκρίνει την, τον κανονισμό αυτό ήδη από το Σεπτέμβριο. Πέναμε τώρα σε ένα άλλο διεθνές όργανο που είναι η Επιτροπή για τους ε, γενετικούς Πόρους ως ό,τι αφορά τη γεωργία και την Επιτροπή της ΦΑΟ. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε προστασία αλλά και αηφόρο χρήση των ε, γενετικών πόρων καθώς και δίκαιη κατανομή των ε, κερδών και των ωφελών από τη χρήση τους. Θα έχουμε τη 13η Σύνοδο της Επιτροπής ε, αυτής που θα γίνει τώρα στη Ρώμη. Εμείς θα ολοκληρώσουμε τις προπαρασκευαστικές εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χάρη στην πολύ καλή προσπάθεια της προηγούμενης Προεδρίας της Ουγγρικής. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα αφιστούμε προσπαθειών προκειμένου να συνεχίσουμε τις ε, εργασίες που ξεκίνησαν σε συνεργασία φυσικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε αν μπορέσουμε αν καταφέρουμε να τις εκπαιρεώσουμε στα πλαίσια της ε, ε, Πολωνικής Προεδρίας. Ε, αν δεν τα καταφέρουμε, τουλάχιστον ε, να προχωρήσουμε τις εργασίες σε μεγάλο βαθμό, ώστε να ολοκληρωθούν το 2012. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Ε, Κύριε Πουκέ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση του προγράμματος της Πολωνικής Προεδρίας. Πρέπει να πω πως έχετε ένα πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο με πολλά θέματα γεωργία, δασοκομεία, αλληλεία σημαντικό κομμάτι για την πολιτική της βιοποικιλότητας μεγάλο θέμα για την οικονομία και την προστασία του κλίματος το είπατε όλα τα μεγάλα θέματα είναι στο δικό σας χαρτοφυλάκιο. Και πράγματι η Πολωνία να προσφέρει πολλά στην Ευρώπη, όπως και η Επιτροπή σας λέει ο κύριος Σαββίτσκι, πράγματι όπως και η Επιτροπή μας, τα μεγάλα αυτά θέματα, προστασία του κλίματος, περιβάλλοντος, βιοπικιλότητας, ε, είναι τα θέματα του 21ου αιώνα. Ακούσαμε το πρόγραμμά σας, η Πολωνία έχει πολλά να προσφέρει, έχετε θαυμάσια τοπία που υπάρχει ακόμα βιοπικιλότητα και μπορείτε να το εξάγετε κιόλα. Αυτή την εμπειρία αυτή σε ολόκληρη την Ευρώπη αναφέρετε τα δάση. Υπάρχουν και πολύ καλά παραδείγματα στην Πολωνία αηφόρου δασοκομείας που πρέπει να γίνει αρχή σε ολόκληρη την Ένωση γιατί έτσι θα έχουμε πολλά, πολλά πλεονεκτήματα. Ξέρω πως βεβαίως σας ενδιαφέρει και η γεωργική πολιτική και η μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Εδώ έχουμε τη γεωργική πολιτική, την, την Επιτροπή την δική μας ε, η οποία συμφώνησε ο πρώτος πυλώνας να πάρει μια, μια πράσινη κατεύθυνση και να δίνονται επιδοτήσεις ε, για τις επιδόσεις ε, και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος η Γεωργία. Και ελπίζουμε να το υποστήριξει αυτό η Προεδρία, γιατί εκεί προς εκεί πρέπει να πάμε. Αναφέρα την Αλία. Εκεί, στο παρελθόν, είχαμε πολλές συζητήσεις υπεραλλιεύουμε, πολλά είδη κινδυνεύουν και ασχοληθήκαμε ειδικά με κάποια με τον τόνο ο οποίος κινδυνεύει με εξαφάνιση και συζητούσαμε το πώς μπορούμε να σώσουμε αυτό το είδος και άλλα, και ψάρια. Και βέβαια αυτό ανήκει γενικότερα στην πολιτική γεωργίας. Είναι σε τεχνολογίες στη γεωργία απασχολούν την Επιτροπή μας. Έχουμε τα νανοηλικά στα τρόφιμα, τα οποία προστίθενται. Ε, εκεί θέμε να ξέρουμε τι συνέπειες έχει αυτό για το ανθρώπινο σώμα και την υγεία. Στον δε κανονισμό νέων τροφίμων συμφωνούσαμε με το Συμβούλιο πως πρέπει να υπάρχει μια σήμανση για να ξέρει πότε ε, υπάρχουν νάνο υλικά μες στο φαΐ ο καταναλωτής. Δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε για, την, για τον κλονισμό των ζώων, την κλονοποίηση Θα δούμε τι πρόταση θα καταθέσει η Κομισιόν στο τέλος του έτους. Εμείς θέλουμε μια νέα πρόταση. Επιτάπητος βεβαίως υπάρχει και ο νόμος περί γενετικής τεχνολογίας. Ε, το Κοινοβούλιο συμμετείχε. Πάμε προς μια επανεθνικοποίηση αυτού του τομέα γιατί δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή θέση και κάθε χώρα θα αποφασίσει από μόνη της αν θα καλλιεργήσει τέτοιους οργανισμούς ή όχι. Και θα θέλαμε να το δούμε αυτό, να λειτουργεί και να γίνει νόμος. Και όμως μπορεί να το ολοκληρώσει αυτό η Προεδρία σας. Ωραία, ε, υπάρχουν και πολλά ακόμα θέματα. Διάβασα επίσης πως ε, τα άλογα πλέον δεν θα τα μαρκάρουν με το σίδερο όπως κάναν παλιά, αλλά θα τους βάζουν ένα τσιπάκι. για να μπορούν να τα αναγνωρίζουν. Είδατε πρόοδος και για τα ζώα, γιατί πονάει και το καημένο το ζώο. Äh, Σας ευχαριστώ λοιπόν. Λοιπόν, ο Ρίχαρτ Τζέμπερ θα κάνει πρώτες ερωτήσεις. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Αναφέρατε τα διάφορα θέματα που θέλει να επεξεργαστεί η Πολωνική Προεδρία. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν αυτό το οποίο ανέφερε και ο Πρόεδρος, ε, οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, που ξέρετε πως ε, το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της ενίσχυσης επικουρικότητας και η δική μου ερμηνεία είναι πως ε, ο κόσμος στην Ευρώπη θα αποφασίσει μόνος του εάν θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα πράγματα στην επικράτεια ενός κράτους ή όχι. Αν θα φυτευτούν για την ακρίβεια. Τι σκοπεύετε για να ξεμπλοκάρει αυτή η δύσκολη κατάσταση στο Συμβούλιο. Ξέρετε πως υπάρχει μια μειοψηφία που μπλοκάρει. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να ε, οδηγηθούμε στην ενίσχυση της επικουρικότητας, όπως είπα. Δεύτερο θέμα, οπωσδήποτε, που μας απασχολεί είναι ασφάλεια των τροφίμων. Ξέρετε πως ανεβαίνουν οι τιμές των τροφίμων και νομίζω εδώ πέρα πως η κοινή γεωργική πολιτική και η κοινή πολιτική αλληλείας είναι σημαντικό κομμάτι. Βεβαίως δεν παίζει τόσο πολύ στα μέσα όπως η κοινή γεωργική πολιτική, αλλά εάν δει κανείς τις πρωτεΐνες και ξέρουμε πως πάρα πολλά είδη υπεραλλιεύονται και ξέρετε πως τα κράτη εκείνα μέλη τα οποία έχουν μεγάλους αλληλευτικούς τόλους είναι κατά της μείωσης των ποσοστώσεων ενώ άλλα κράτη που δεν έχουν τέτοιον κλάδο είναι αδιάφορα. Τι σκοπεύετε να κάνετε ε, για να υπάρχει η δυνατότητα μακροπρόθεσμα να ψαρεύουμε τέλος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Νομίζω είδατε πως ε, στη ΣΥΠΑ ε, έχουμε πλέον μεγαλύτερη κατανάλωση δημητριακών ε, για παραγωγή ενέργειας από ότι για τρόφιμα. Δεν μπορεί να έχουμε και εδώ την ίδια κατάσταση. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να προωθηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά να μην υπάρχει ανταγωνισμός με τα τρόφιμα. Ευχαριστούμε, Άντρες Πυρίλο, που ήταν βεβαίως ε, εισηγητής και για τους χυμούς φρούτων και θα μας ρωτήσει πώς η ζάχαρη επιτρέπεται να έχουν χυμή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για την παρουσίασή σας, όπως είπε και ο κύριος Λένιν. Εργάζομαι για την τροποποίηση της οδηγίας ε, για τους ε, χυμούς από ε, φρούτα και θέλω να κάνω μια σχετική ερώτηση και μια διευκρίνηση. Η ερώτηση, τι πιστεύετε εσείς για την εφαρμογή του Κόντεξ Ελιμεντάριους και ποια είναι η θέση σας σε σχέση ε, με την εφαρμογή του. Είναι, δεν, ε, είναι η αλήθεια ότι δεν μας δεσμεύει αλλά ουσιαστικά διέπει την διατροφική πρακτική στην Ευρώπη και στον κόσμο. Όταν ε, αρχίσαμε να συζητούμε την τροφή της οδηγίας ουσιαστικά αντιμετωπίσαμε αφενός το τι πιστεύουν τα κράτη και τι επιτρέπει επιτρέπουν ε, στις εισαγωγές ε, σε ό,τι αφορά την οξύτητα των προϊόντων και ε, επίσης αν απαιτούσαμε την ίδια προϋπόθεση, τις ίδιες προϋποθέσεις για όλα τα προϊόντα τότε μπορεί να είχαμε πρόβλημα στον ΠΟΕ, προσφυγή στον ΠΟΕ κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως αν εφαρμόσουμε τον κότεξ σε ευρωπαϊκά προϊόντα, παραδείγματο χάρη για την ε, προσθήκη χυμού μαντερινιού σε ορισμένα προϊόντα, λέμε ότι αυτό δεν ισχύει. Έχουμε λοιπόν διτή εφαρμογή. Αν ε, ε, έχουμε, έχουμε μάλλον ορισμένα προϊόντα για τον οποία εφαρμόζουμε τον κόντεξ και άλλα προϊόντα για τον οποία δεν εφαρμόζουμε τον κόντεξ, είναι πιο περιοριστικό. Έτσι λοιπόν θέλω να σα ρωτήσω τι πιστεύετε για την εφαρμογή ε, ή πώ πρέπει τέλο πάντων να τηρούμε αυτό τον κανόνα και μια διευκρίνηση που δεν έχει να κάνει με αυτό. Ε, αναφερθήκατε στα δάση και κατάλαβα ότι εσείς ε, θέλετε κάποια στιγμή να έχουμε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία ή μια οδηγία για τα δάση που να σέβεται και την ποικιλομορφία των ε, διάφορων ειδών του ευρωπαϊκού ε, δάσους. Αλλά αν δεν κάνει αυτό τουλάχιστον εσείς θέλετε να τίθεται ορισμένοι ελάχιστοι κανόνες, δηλαδή να έχουμε ένα κοινό κανόνα που να περιλαμβάνει τα είδη της προστασίας, τα είδη της ε, δασοκομείας ε, και πώς θα γίνονται οι επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν κατάλαβα καλά, εσείς ήσασταν είστε υπέρ κάποια στιγμή να έχουμε μια τέτοια ευρωπαϊκή οδηγία για τα δάση, έτσι ώστε να έχουμε κάποια ε, κοινά ελάχιστα σε ό,τι αφορά την προστασία των δασών και να καλύπτουμε πλήρως τον όρο δάση, ευρωπαϊκά δάση. Σας ευχαριστώ. Thank Κυρία Ντεμπρίν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον Υπουργό που παρευρίσκεται εδώ σήμερα και που μοιράστηκε τις σκέψεις του μαζί μας. Επίσης, χάρηκα πολύ που άκουσα τα σχολεία του Υπουργού, κυρίως για τα δάση, καθώς ήμουν σκιώδης ε, εισηγήτρια για αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση. Επομένως, θα ήθελα να ακούσω περισσότερες λεπτομέρειες ε, για όσα ε, θεωρείτε θετικά και θεωρείτε ότι μπορείτε να προωθήσετε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Ε, έρχομαι από την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Επομένως, ε, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλήσατε για την απλουστευμένη ταυτοποίηση των εγωπροβάτων. Όμως, ε, για την μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής. Ε, είπατε ότι υπάρχει ρεαλιστική προσέγγιση προς αυτό. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν ε, κάτι για τα κίνητρα στους γεωργούς για να έχουν πιο ορθή διαχείριση των γεών και έναν ισχυρό δεύτερο πυλώνα υπήρχε και ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γι' αυτό και σε ό,τι αφορά τον πρώτο πυλώνα και την κατευθύνση του πρασινίσματος ε, μιλήσατε γι' αυτό και στις προεδρικές σας κύριε Υπουργέ. Πώς ε, βλέπετε να κινούνται τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση στις συζητήσεις που έχετε με τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά είτε τη θέσπιση δράσεων ε, είτε την ευελιξία σε επίπεδο κρατών μελών και ε, πιστεύετε ε, ότι πέρα από το ποια κατεύθυνση θα αποφασιστεί, πιστεύετε ότι θα μπορούν ε, να υπάρχουν σαφώς προσδιορισμένες και εύκολα μετρήσιμες πράξεις χωρίς να έχουμε υπερβολική γραφειοκρατία και τελικά να καταλήξουμε στα αποτελέσματα τα οποία όλοι προσδοκούμε. Ευχαριστώ, Καρλ Χάιντς Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Χάρηκα πολύ με αυτά που είπατε. Εγώ δεν θα ρωτήσω για τον προπολογισμό. Εμένα με ενδιαφέρει το πώς ε, θα μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτή την ε, μεγάλη συγκέντρωση του εμπορίου στα χέρια ολίγων. Παραδείγματος χάρη στη Γερμανία υπάρχουν μόνο 8 άτομα τα οποία αγοράζουν ε, ε, χοιρινό κρέας. Δεν υπάρχει πλέον αγορά, μιλάμε για ένα καρτέλ και στο τέλος θα καταλήξουμε να δούμε πως το γάλα θα είναι φτηνότερο από το μεταλλικό νερό. Τι θα γίνει με αυτή την ε, υπόθεση. Κατόπιν για το κλίμα εντάξει και τα λοιπά, για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Δεν ξέρω αν θα ήθελα αυτό το οποίο θέλει ο Ρίχαρτ Τζέμπερ, μια επανεθνικοποίηση. Εγώ ζω 9 χιλιόμετρα από τα Ολλανδικά σύνορα και οι Ολλανδοί έχουν επιτρέψει εκεί πέρα γενετικά τροποποιημένους ε, οργανισμούς. Ε, δεν υπάρχουν πλέον σύνορα και έρχεται να μάξει με ζωοτροφή στο Ρήνο όπου ζω εγώ και δεν δηλώνει κανείς, δεν υπάρχει πουθενά στα έγγραφα το εάν αυτή η τροφή των γουρουνιών έχει μέσα γενετικά ε, τροποποιημένα τρόφιμα ή όχι. Τα δίνει εκεί πέρα στη Γερμανία και ανακαλύπτει ο Γερμανός κτηνοτρόφος στο σφαγείο πως κάπου υπήρχαν στην όλη αυτή η διαδικασία ε, γενετικά τροποποιημένοι αυτη διαδικασια γενετικα τροποποιημενοι οργανισμοι Το πρόβλημα θα μεγαλώσει λοιπόν πάρα πολύ με αυτή την κατάσταση. Οπότε, ε, ξέρετε, το θέμα είναι, γιατί έχω και συνεργάτη σε πολωνική επιχείρηση, τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Ευχαριστούμε, Καλχάνης Φλόρεντς. Ε, πρέπει να προσέχει κανείς από πού προέρχεται, από πού αγοράζει τις ζωοτροφές και τα υλικά. Δεν είναι απλό. Ε, θα σας απαντήσει ο κύριος Υπουργός. Βιτόριο Πρόντι, λοιπόν. Ε, ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ που παρευρίσκεστε εδώ. Εγώ θέλω συγκεκριμένα να επιμείνω στα ε, απόβλητα από τη γεωργία και από τη δασοκομεία και στην ε, δυνατότητα ε, να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο έτσι ώστε να μετατρέψουμε αυτή την βιομάζα σε αέριο στα υπολείμματα λοιπόν από τη Γεωργία για τη δασοκομεία. Έτσι λοιπόν ε, να βρούμε ένα τρόπο για να αυξήσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα φενός και φετέρου μέσω αυτής ε, της χρήσης των νεώσιμων πηγών ε, να βρούμε και τους πόρους για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, κάτι που είναι απαραίτητο σε όλη την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν ε, βλέπω ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία αυτού του τομέα. μπορούμε να πούμε, παίρνουμε το σχάρι, ότι ένας τόνος ε, ξηρής βιομάζας ε, μας δίνει περίπου χίλια κυβικά μέτρα υδρογόνου μέσω της πυρόλησης. Δεν είναι αμεληταίο λοιπόν σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα εγώ νομίζω ότι αν δούμε και τι συμβαίνει στην Ιταλία, μόνο από αυτά τα υπολείμματα των δασών και της γεωργίας εμείς ε, μπορούμε να καλύψουμε το 1 τρίτο των αναγκών μας αέριο. Όμως πρέπει να γίνει αυτή η αξιολόγηση ε, και αυτή η αξιοποίηση και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εσείς θεωρείτε ότι μπορείτε να αναλάβετε με τέτοια πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ehm, Ευχαριστούμε, Βιτόριο. Κατόπιν, Αλόης Πέτερλε, ο οποίος είναι μελισσοκόμος αυτός και ασχολείται με τις μέλισσες στην Ευρώπη. Αλόης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν υπάρχει σλοβενική μετάφραση, να μιλήσω αγγλικά. Ευχαριστώ που αναφέρατε και το χόμπι μου, το οποίο γίνεται όλο και πιο απαιτητικό. Ήταν ε, ρομαντικό να είναι κανείς μελισσοκόμος πριν από 20-30 χρόνια, αλλά όχι πια. Ξέρετε σε τι αναφέρομαι. Τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ ε, έχουμε θάνατο των μελισσών ε, σε μεγάλους αριθμούς. Οι μέλισσες είναι κατά την άποψή μου ο καλύτερος δείκτης της ποιότητας του περιβάλλοντος και εμείς υιοθετήσαμε χτες μια γνωμοδότηση για την υγεία των μολυσσών. Ήταν ενδιαφέρον που είδαμε πάνω από 150 τροπολογίες μόνο στη γνωμοδότηση, όχι σε έκθεση. Οπότε γνωρίζουμε το τι συμβαίνει. Και νομίζω πως ακόμα δεν έχει δοθεί προσοχή στο θέμα αυτό, στον δίκτυ ας πούμε. Και νομίζω πως σχετίζεται με το πρώτο μέρος της παρουσίασής σας μιλούσατε για ασφάλεια των τροφίμων. Νομίζω πως χρειάζεται πιο συνολική προσέγγιση και νομίζω πως μέσω των μελισσών μπορούμε να δούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Πρέπει να δούμε το πλαίσιο. Το περιβάλλον δηλαδή. Και χρειάζεται μία γενικότερη προσέγγιση, όχι απλά κάποιες βελτιώσεις. Δεν θα τις έλεγα διακοσμητικές, αλλά πρέπει να ασχοληθούν πολύ περισσότερο με το ζήτημα της χημείας ε, στη γεωργία κτλ. <laughs> In that respect, but I think that this development... Ε, νομίζω λοιπόν πως αυτές οι εξελίξεις ε, των τελευταίων ετών είναι πολύ σημαντικές και απαιτούν πολύ περισσότερη προσοχή και ξέρω πως και οι Πολωνοί μελισσοκόμοι το γνωρίζουν το θέμα. Yeah. Uh, uh- ναι, το πολωνικό μέλι είναι λιχουδιά και θέλουμε μέλι και στο μέλλον. Και είναι καλός δείκτης για την ποιότητα του περιβάλλοντος μέλισσες. Λοιπόν, Καρίν Κάλενμπαχ. Και εγώ θέλω να αναφερθώ στο ίδιο. Χάρηκα για το ότι χτες έγινε δεκτή η τροπολογία μου που αναφέρθηκε ε, βεβαίως πως ε, μάλλον ε, τα εντομοκτώνα και οι γενετικά τροπημένοι οργανισμοί έχουν κάποια επίδραση. Και έρχομαι στους γενετικά τροπημένους οργανισμούς, όπου βρίσκομαι πολύ πιο κοντά στον Ρίχιαρντ από ότι στον κύριο Φλόρεντς. Ε, καθυστέρησα λίγο και δεν άκουσα όλες τις δηλώσεις σας, αλλά Ξέρετε πως ε, συζητάνε στην Επιτροπή Γεωργίας το πλαφόν στις πληρωμές και θα με ενδιέφερε του πρώτου πυλώνα. και τη μετάβαση στον ε, δεύτερο. Οπότε με ενδιαφέρει ως μέλος και της Επιτροπής Περιβάλλοντος το ποια μέσα θα διατεθούν στον δεύτερο πυλώνα. Μάλιστα κύριε Υπουργέ, πολλές ερωτήσεις ενδιαφέρουσες Αναμένουμε απαντήσει, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση όντω. και εμείς και για τη Γεωργία και για την Αλία δεν καταφέρουμε να έχουμε ε, πάντα δεκαετή προοπτική και μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Θα πρέπει όμως να ασχοληθούμε πια πολύ σοβαρά με την κυνηγερική πολιτική και πολύ διαπιστώνουμε ότι η κοινή γεωργική πολιτική είχε και πολλά μειονεκτήματα και έκανε και πολλά κακά και αυτά θα πρέπει να τα διορθώσουμε. Μία Ευρωβουλευτής μας υπενθύμησα ότι είπα ότι εγώ έχω μια ρεαλιστική προσέγγιση για την ε, κοινή γεωρική πολιτική. Όχι. Εγώ έχω μια πολύ απαιτητική προσέγγιση για την κοινή γεωρική πολιτική και περιμένω πραγματικά ε, μια ρηξικέλευτη και βαθιά μεταρρύθμιση. Η ρεαλιστική προσέγγιση οθετεί κυρίως η Επιτροπή Γεωργίας που ανταποκρίνεται και στην κρατούσα γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και νομίζω ότι η ρεαλιστική προσέγγιση οθετεί και το Συμβούλιο. Α, τώρα, σε ό,τι φορά τις μέλισσες της συνύπαρξης των διαφόρων ειδών στο περιβάλλον, το θέμα των χημικών προϊόντων. Τα πρώτα 20 χρόνια της κοινή γεωρικής πολιτικής ε, ε, διαπιστώσαμε μια εντατικοποίηση της παραγωγής, ε, μαζική χρήση χημικών προϊόντων και τώρα αρχίζουμε και προβληματιζόμαστε. Πού χάθηκε η βιοπικιλότητα της Ευρώπης, τι ζημιές προκάλεσε στην Ευρώπη μόνο μονοκαλλιέργεια. Πώς θα εμπλουτίσουμε και πάλι το έδαφος. Και τι είναι τελικά το έδαφος. Είναι απλώς ένα, το, ένα υπόθεμα της παραγωγής ή είναι και πραγματικό φυτόριο της βιοπικιλότητας. Ποιο είναι ο ρόλος του εδάφους. Και σε αυτά τα ζητήματα Έχουμε να πούμε πολλά στα πλαίσια τη γεωργική πολιτική. Και μάλιστα το φθινόπωρο θα διοργανωθεί στι Βρυξέλλε μία διάσκεψη με θέμα την βιολογική ανανέωση του εδάφους και τον εμπλουτισμό του εδάφους. Και βλέπουμε ότι σε ό,τι αφορά τη χρήση των λιπασμάτων, στην Κίνα για παράδειγμα, και πόσο ε, αλλάζει το έδαφος εξαιτίας αυτών, όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Γι' αυτό και η μεταρρύθμιση της κοινή γεωρικής πολιτικής ε, δεν μπορεί να ε, ερμηνευθεί μόνο από οικονομική άποψη. Βέβαια, δυστυχώς, το 90% των συζητήσεων στην Ευρώπη περιορίζονται στα οικονομικά ζητήματα και στη σύγκριση. Ποιος κερδίζει, ποιος χάνει, ποιος δίνει, ποιος παίρνει. Πιστεύω όμως ότι εμείς ως Ευρωπαίοι δεν βρήκαμε ακόμη το θάρρος να εξετάσουμε τη γεωργία με ευρωπαϊκό και πιο σφαιρικό και ολοκληρωμένο τρόπο. Αναφέρθηκε και το θέμα των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. Είναι ένα ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής. Εγώ βλέπω τεράστια διαφορά και διάσταση απόψεων. Ε, η ευρωπαϊκή επιστήμη δεν μας δίνει τεκμηριωμένα και βάσιμα επιχειρήματα για να μπορούμε να κάνουμε σύγκριση ε, το, της χρήσης ή μη χρήσης των γενετικών τροποποιημένων οργανισμό και τι επιπτώσεις έχουν. Δεν είμαστε σε θέση να πούμε σήμερα αν και κατά πόσο γενετικώ τροποποιημένοι οργανισμοί ε, απειλούν την βιοπικιλότητα. Υπάρχουν φημολογίες ότι την απειλούν. Εμείς φυσικά θέλουμε να προφυλάξουμε τη βιοπικιλότητα και μερικές φορές μπλοκάρουμε για αυτό το λόγο την καλλιέργεια γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στην Ευρώπη. Αλλά έτσι ε, είπαμε να εκχωρήσουμε τις αποφάσεις στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Και πολύ σωστά ο κύριος Φλόρεντς ε, ε, προβληματίστηκε ε, τι θα γίνει στην περίπτωση των παραμεθόριων περιοχών όταν μια χώρα υιοθετεί διαφορετική προσέγγιση για τους γενετικώς ε, τροποποιημένους οργανισμούς από την γειτονική της. Το ίδιο συμβαίνει με τη Τσεχία και την Πολωνία που είναι γειτονικέ χώρες. Αν μια χώρα επιτρέπει και μια απαγορεύει. Αλλά μερικές φορές με τέτοιες άκαμπτες απόψεις ε, εμποδίζουμε το άνοιγμα της Ευρώπης. Εγώ χρειάζομαι βάσιμα επιστημονικά, βιολογικά, οικονομικά επιχειρήματα. Εμείς στην Ευρώπη λέμε δεν θα καλλιεργήσουμε γενετικώ τροποποιημένους οργανισμούς και φυτά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες α πούμε. Απ' την άλλη πολύ ευχαρίστως θα εισαγάγουμε γενετικώ τροποποιημένε ζωοτροφέ από άλλες περιοχές του κόσμου και δεν βάζουμε κανένα φραγμό ε, για την εισαγωγή μεταλλαγμένων τροφίμων από άλλε χώρε, γιατί λέμε ότι ο καταναλωτή έχει το δικαίωμα επιλογή, έχει το δικαίωμα να αγοράσει φθηνά προϊόντα. Λέμε λοιπόν εμεί οι Ευρωπαίοι. Θέλουμε να προφυλάξουμε την ευρωπαϊκή βιοπικιλότητα. Σε πολλές περιοχές της Ευρώπης ε, θα πρέπει να ξαναδημιουργήσουμε την βιοπικιλότητα, γιατί πραγματικά εκεί υπήρξε διαταραχή και απειλή της βιοπικιλότητας. Αλλά θέλω τυφλούμε, γιατί ταυτόχρονα χάρη σε μια φιλελεύθερη προσέγγιση που εθετούμε για την αγορά, λέμε «Α, δεν πειράζει, ας καταστραφεί η βιοπικιλότητα σε άλλες περιοχές του κόσμου, δεν μας ενδιαφέρει». Οι δικές μας επιστησικές ανάγκες, ε, εκτός στην Ευρώπη, ε, έχουμε ε, 300 εκατομμύρια ε, εκτάρια καλλιέργειες για ζωοτροφές που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη. Και το θέμα των γενετικώς τροπημένων οργανισμών δεν θα πρέπει να το εξετάσουμε μόνο σε στενά όρια της δικής μας περιοχής, του Δήμου, της κοινότητας ή του κράτους, αλλά θα πρέπει να το δούμε με πιο σφαιρικό τρόπο. Η προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή στο Συμβούλιο Υπουργών είναι ισορροπημένη, αλλά στη συζήτηση θα πρέπει να προσέξουμε και να μην απομακρυνθούμε από τα επιστημονικά πορίσματα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και να απαιτούμε επιστημονικές τεκμηριωμένες μελέτες για τα θέματα αυτά. Γιατί σίγουρα δεν είμαστε ε, στην Ευρώπη πρωτοπόροι στις βιοτεχνολογίες. Χρειαζόμαστε όμως επιστημονικές μεθόδου, μεθόδους και γνώσεις για το θέμα αυτό και επιχειρήματα. Το ίδιο ισχύει και για την κλωνοποίηση. Στην ε, ευρωπαϊκή και παγκόσμια γεωργία έχουμε τόσο τεράστιο δυναμικό παραγωγής και ανάπτυξης, ώστε μπορούμε για πολλά χρόνια να εξασφαλίσουμε τον επιστηστικό ανεφοδιασμό και στην Ευρώπη και στον κόσμο, χωρίς ε, να χρειαζόμαστε ούτε κλωνοποίηση ούτε γενετικό τροποποιημένο οργανισμό. Αλλά αυτό προϋποθέτει μια πραγματικά κοινή γεωρική πολιτική και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και όχι στενή εθνική ή αμυγός οικονομική προσέγγιση για τη γεωργία. Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε στο ζήτημα της αηφόρου αηλίας, της απώλειας των αποθεμάτων των τόνου. Με ικανοποίηση έμαθα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χάρη στα μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης αποθεμάτων η κατάσταση για τον τόνο είναι κάπως καλύτερη. Και έχουμε όλο και καλύτερες και τελειότερες επιστημονικές μεθόδους για τον έλεγχο των ηχθιαποθεμάτων. Βέβαια, πολλές φορές βλέπουμε ότι οι ίδιοι οι αλείς μερικές φορές ε, δεν, προβλέπουν, ε, δεν, δεν προβαίνουν σε πλήρη ταυτοποίηση και καταχώρηση των και μερικές φορές ε, δεν έχουμε ε, πλήρη στοιχεία. Και το θέμα των απορρίψεων επίσης δεν τα έχουμε διευθετήσει. Πώς θα το χειριστούμε. Γιατί και εκεί έχουμε σημαντικές απώλειες. Και εδώ ανακύπτει το ζήτημα της περιφερειοποίησης ε, της αλίας και έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε τους ίδιες διατάξεις να τις εφαρμόζουμε ε, σε, σε λεκάνες που έχουν τελείως διαφορετική σύσταση, χαρακτηριστικά, ιδιότητες. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τις διαστάσεις, ε, τα αλληλευτικά αποθέματα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη για να δούμε πώς με ορθολογικό τρόπο θα εργαστούμε σε αυτό το πολύμορφο αλληλευτικό περιβάλλον. Το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το επισήμανα και εγώ. Ε, είπα ότι πριν από 100-120 χρόνια η Γεωργία ήταν ενεργειακά αυτάρκης. Το 2007, το 2008 μάλλον, ακούσαμε ότι η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, από τρόφιμα δημιούργησε τεράστιες αναταραχές γιατί ε, η παραγωγή βιοκαυσίμων οδήγησε σε αύξηση των σιτηρών, της τιμής σιτηρών στην Ευρώπη. Βέβαια, είχαμε το αντίθετο. Εγώ διαπίστωσα μείωση κατά 50%. Αν τουλάχιστον ένα τόνο ε, λιγότερα σιτηρά το, δεν, το, δεν τα χρησιμοποιούσαμε γιατί βιοκαύσιμα αλλά για τη βιοεθανόλη, δεν θα είχαμε τέτοια αύξηση. Τελικά μειώθηκαν οι τιμές των σιτηρών, παρόλο που είχαμε ίδια παραγωγή βιοκαυσίμων. Ο συναγερμός λοιπόν αυτό ήταν ανεδαφικός. Περισσότερο για κερδοσκοπία πρόκειται παρά για πρόβλημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα πρέπει να δούμε τι ποσότητα τροφίμων θα την τι ε, τμήμα των σιτηρών θα το αφιερώσουμε στην παραγωγή των βιοκαυσίμων. Θα πρέπει να δούμε και το θέμα της ε, ασφάλειας των τροφίμων. Επίσης υπάρχουν, έχουμε πολλά οργανικά απόβλητα και εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σωστή αξιοποίηση. Έχουμε την ηλιακή ενέργεια, την αιωλική ενέργεια. Έχουμε πάρα πολλά θέματα εδώ για τις ανανεώσιμες πηγές που θα πρέπει να τα εξετάσουμε και να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες των πιο προηγμένων χωρών στις τεχνολογίες αυτές, ώστε να κάνουμε μια σωστή διαχείριση των πηγών αυτών και του περιβάλλοντος. Υπάρχει και το θέμα, πολύ σημαντικό θέμα, της βιομάζας των δασών. Δεν θα ήθελα σήμερα η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από τη βιομάζα να αποτελέσει λόγο ή πρόσχημα για την ε, ε λαιλασία των δασών. Δεν θα πρέπει να πέσουν ε, τα δάση θύμα στο βωμό των δασών. Γιατί μερικές φορές ε, υπάρχει πειρασμός ε, λόγω της κερδοφορίας να χρησιμοποιούν όχι μόνο τα απόβλητα των δασών, αλλά να χρησιμοποιηθεί και η υλοτομία, το ξύλο. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει πραγματικά σε ελαφυραγώγηση των δασών. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε και να είμαστε πολύ απαιτητικοί και πολύ περιοριστικοί. Δεν μπορούμε να θυσιάσουμε τα δάση μας και στο βωμό της ανανεώσιμης ενέργειας να καταστρέψουμε το φυσικό μας περιβάλλον και να αποψηλώσουμε τα δάση μας. Κάτι τέτοιο νομίζω είναι απαράδεκτο. Συμφωνώ και με τον Ευρωβουλευτή που είπε ότι οι μέλισσες είναι ένας φυσικός ε, δείκτης της ποιότητας του περιβάλλοντος. Έχω όμως την εντύπωση ότι πολλές φορές τα προβλήματα των μελισσοκόμων σε μεγάλο βαθμό ε, για τα προβλήματα μάλλον των μελισσοκόμων σε μεγάλο βαθμό κατηγορούμε τους γεωργούς και στην ε, Πολωνία έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Γι' αυτό και κάνουμε μελέτες και προσπαθούμε να διαγνώσουμε τις αιτίε της μεγάλης θνησιμότητας των μελισσών. Γιατί πραγματικά έχουμε υπερβολική θνησιμότητα των μελισσών. Προσπαθούμε να δούμε αν τα φυτοφάρμακα είναι η αιτία σε μεγάλο βαθμό αυτής της θνησιμότητας. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που διαταράσσουν το φυσικό περιβάλλον και άρα συμβάλλουν στην αύξηση της θρησιμότητας των μελισσών. Δεν είναι υπεύθυνοι για όλα οι γεωργοί. Γι' αυτό θα πρέπει να εντείνουμε και τις μελέτες και τις επιστημονικές έρευνες και να προστατεύσουμε το περιβάλλον όχι μόνο μέσω της γεωργίας αλλά μέσω και της οικονομικής διαχείρισης που κάνουμε και άλλων κλάδων. Ένα άλλο θέμα που επισημάθηκε ήταν η χρήση της ζάχαρης και το θέμα του κόντεξ alimentariums. Για τους ε, παραγωγούς ε, τροφίμων στην Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια, για τους ε, Ευρωπαίους παραγωγούς τροφίμων, τα τελευταία χρόνια επιβάλαμε και απαιτήσαμε πολύ ψηλές προδιαγραφές είχαμε τεράστιες απαιτήσεις. Και αυτή τη στιγμή στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου αλλά και σε διμερείς και τριμερείς διαπραγματεύσεις και στις συμφωνίες με το Μερκοσούρ έχουν προχωρήσει πολύ οι συζητήσεις. Όλες οι περιοχές του κόσμου περιμένουν ε, από την ευρωπαϊκή αγορά ε, να συντηρηθούν οι γεωργοί όλου του κόσμου από τις αγορές των Ευρωπαίων καταναλωτών. Προσοχή όμως, έχουμε υψηλές απαιτήσει και προδιαγραφές για τους δικούς μας παραγωγούς, γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να εξασφαλίσουμε την ευημερία των ζώων. Αλλά δεν μπορούμε ταυτόχρονα στην Ευρώπη, εμείς έχουμε τόσο υψηλές απαιτήσει από τους δικούς μας παραγωγούς και ταυτόχρονα να αφήνουμε ξέφραγο μπέλη, να ανοίγουμε διάπλατα τις πόρτες μας σε προϊόντα και να εισαγάγουμε προϊόντα που δεν τηρούν αυτές τις προδιαγραφές. Το ίδιο ισχύει και για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε και να προφυλάξουμε τη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη, γιατί να μην προφυλάξουμε τη βιοποικιλότητα και των άλλων περιοχών του κόσμου, γιατί και σε άλλες περιοχές του κόσμου χρειαζόμαστε τη βιοποικιλότητα. Το ίδιο ισχύει και για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων. Ίδιες απαιτήσει θα πρέπει να έχουμε και για τους εταίρους μα και όχι μόνο να τι επιβάλλουμε εντός της Ευρώπης η Ευρωβουλευτή μίλησε για το θέμα του πρασινίσματος εντός εισαγωγικών. Πολύ συχνά στι συζητήσεις μερικές φορές ε, αποδεσμευόμαστε από προηγούμενες ε, λύσεις και αποφάσεις. Το 2003, όταν έγινε η αποδέσμευση των ενισχύσεων από την παραγωγή, ε, ήταν καλή η λύση γιατί έδωσε στους γεωργούς μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής με προσανατολισμό προς την αγορά και ανάλογα με τις πληροφορίες που ανάλαβαν με την αγορά τελικά υιοθετήσαμε μία αρχή της ε, αμοιβές ε, ωφέλειας κατά κάποιο τρόπο δηλαδή θα έπρεπε να εξηγήσουμε στον καταναλωτή ότι επιβάλλαμε στους γεωργούς πολύ ε, απαιτητικές προδιαγραφές. Κάτι που δημιούργησε υποχρέσεις ε, ε, για 6-7 γενιές γεωργών. Παρ' όλα αυτά, ξε... υιοθετήσαμε αυτές τις διατάξεις, ε, μοιράσαμε χειρίδες στους γεωργούς και τώρα ε, κάνουμε ένα αυστηρό έλεγχο κατά πόσο τα, τα βιβλιάρια τους θα συμπληρώνουν οι γεωργοί και αν τηρούν αυτές τις νομοθετικές διατάξεις. Και στα πλαίσια αυτών των ε, διατάξεων έχουμε και δεύτερο τμήμα που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένες υποχρεώσεις ε, που φέρουν οι γεωργοί για την προστασία του περιβάλλοντος και αναφέρονται όλα αυτά πολύ λεπτομεριακά. Επιπλέον έχουμε και οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Φαίνεται τώρα ότι αν ε, ε, καταρτήσουμε ένα χάρτη με την υλοποίηση όλων αυτών των υποχρεώσεων, για να δούμε πού εφαρμόζονται, σε πολλές ε, περιοχές αυτός ο χάρτης ήταν κενός. Εξαιτίας της μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις. Τώρα, θα πρέπει στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα, που κανονικά θα πρέπει να είναι ο πυλώνας αποζημίωσης για την αυστηρή συμμόρφωση με τους κανόνες, θα πρέπει αυτό να το τηρήσουμε ώστε όλες αυτές οι διατάξεις που υιοθετήσαμε να γίνουν σεβαστές, να εφαρμόζονται στην πράξη. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, ο Ευρωπαίος Γεωργός που θα εμπίπτει στον πρώτο πυλώνα θα είναι ο πραγματικά φιλοπεριβαλλοντικός Γεωργός, ο πράσινος Γεωργός. Και φυσικά θα πρέπει να εμπλουτίσουμε την προσπάθεια πρασινίσματος γεωργίας, αλλά όχι με αρχή της υποχρέωσης για όλους. Ο πρώτος πυλώνας είναι υποχρεωτικός και αυτός είναι ο πιο πράσινος γεωργός, ο πιο φιλοπεριβαλλοντικός. Αν θέλουμε να είμαστε πιο απαιτητικοί, στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα, με ενάυσματα, όχι με επιβολή υποχρεώσεων, με ενάυσματα, με κίνητρα, πενταετή, με πενταετή, εξαετή, πολυετή σχέδια με δημοσιονομική υποστήριξη να συνεχίσουν την περαιτέρω, το περαιτέρω πρασίνισμα της Γεωργίας. Όχι όμως με επιβολή υποχρεώσεων όπως στον πρώτο πυλώνα, αλλά με παροχή εναυσμάτων και κινήτρων στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα. Συχνά επαναλαμβάνω ότι αν η Ευρωπαϊκή Γεωργία επικεντρωθεί στις άμεσες ενισχύσεις, στις άμεσες πληρωμές για να επιφέρει μια οικονομική σταθεροποίηση, αυτή η γεωργία θα είναι αμυντική, συντηρητική, προσανατολισμένη μόνο προς την παραγωγή. Αν στο δεύτερο πυλώνα δώσουμε έμφαση στον εταιρισμό, στην καινοτομία, στην ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα, με ένα σύστημα εναυσμάτων και κινήτρων για τους πιο φιλοπε... φιλοπεριβαλλοντικούς γεωργούς, τότε θα καταφέρουμε να απελευθερώσουμε τη γεωργία από αυτή τη στασιμότητα του πρώτου πυλώνα. Είπε ο Αλμπερντές πώς για 30 χρόνια είχαμε αύξηση της γεωργικής παραγωγής σε άλλες περιοχές του κόσμου και όχι στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη έχουμε μία στασιμότητα. Ενώ το αναπτυξιακό δυναμικό της γεωργίας, χωρίς καν να προσφεύγουμε σε γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, χωρίς καν να χρειαζόμαστε την κλωνοποίηση, Χωρί υπερβολική χρήση λοιπασμάτων και χημικών προϊόντων, το αναπτυξιακό και το παραγωγικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Γεωργίας δυστυχώ βρίσκεται ακόμη σε λανθάνουσα κατάσταση. Έχει μείνει αναξιοποίητο. Θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε περισσότερο. Βαθύτερο πρασίνισμα λοιπόν στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα και εφαρμογή υποχρεώσεων στα πλαίσια των υποχρεωτικών διατάξεων του πρώτου πυλώνα. Ένα άλλο ερώτημα αφορά την απειλή και τα προβλήματα που δημιούργησε το κολοβακτηρίδιο, ασχερίδια κόλλη. Το σύστημα έγκυρης προειδοποίησης φαίνεται ότι δυστυχώς δεν λειτουργεί ακόμη σωστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λένε οι πολέμοι του. Κατά τη γνώμη μου το σύστημα αυτό λειτουργεί σωστά και τα περιφερειακά υγειονομικά συστήματα ε, Εκεί ήταν που υπήρχε το πρόβλημα, όχι στο ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Τα περιφερειακά συστήματα μας απογοήτευσαν. Θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τα εθνικά ελεγκτικά μας συστήματα και υγειονομικά συστήματα, αλλά δεν αρκεί αυτό. Θα πρέπει να εθωτήσουμε διαφορετική αντίληψη για την παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη και στον κόσμο. Γιατί εκβιομηχανίσαμε τη γεωργία και προσπαθήσαμε να αυξήσουμε την παραγωγή νομίζοντας ότι ξεχνώντας ότι το καλύτερο προϊόν είναι αυτό που παράγεται κοντά στο χώρο πώλησης. Αυτό θα είναι και το πιο φθηνό. Και θα είναι και το πιο ποιοτικό και το θα δημιουργήσει τέτοιες απειλές όπως η βιομηχανική παραγωγή. Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις του κυρίου Τσόλος, για την ε, νέα γεωρική πολιτική απέναντι στους νέους παραγωγούς ε, ε, ως προς τη μεταποίηση των προϊόντων, ως προς τις άμεσες πωλήσει. Όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά. Να εξετάσουμε τη μικροαγορά, της, την παραγωγή που γίνεται κοντά στο χώρο πώλησης από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Ντόπια προϊόντα. Νομίζω ότι έτσι και τις απειλές θα περιορίσουμε και την προστασία του περιβάλλοντος θα εξασφαλίσουμε. Γιατί να πρέπει ο παραγωγός να στέλνει στα 300 χιλιόμετρα στο εργοστάσιο ε, να μεταποιηθεί το προϊόν του και να ε, επιστρέψει να το πουλήσει κοντά στην περιοχή του ή να το πουλήσει ακόμη πιο μακριά. Θα πρέπει να μειώσουμε την απόσταση αυτής της αλυσίδας. Αυτό θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα που θα είναι ο πιο ενεργός, ο πυλώνας που θα είναι στραμμένος προς την ανάπτυξη, την καινοτομία και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της τροφικής αλυσίδας, και εκεί θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να μην επαναλαμβάνω αυτό που κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια, ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των γεωργών, να τους δώσουμε ευκαιρίες να οργανωθούν καλύτερα, να στηρίξουμε τις οργανώσεις γεωργών. Θα πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο να, να περιορίσουμε την ε, έλλειψη εντιμότητας που υπάρχει μερικές φορές στο εμπόριο. Υπάρχει εσχροκέρδεια στο εμπόριο. Γιατί μερικές φορές στο εμπόριο επικρατούν λίγοι πολυεθνικοί όμιλοι και αυτό το λιγοπόλιο επιβάλλει τους κανόνες του και στους γεωργούς και στους μεταπίτες. Θα πρέπει λοιπόν και αυτό το θέμα να το εξετάσουμε. Να δούμε τι κανόνες θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε. Αναφέρθηκε και το ζήτημα της ευημερία των ζώων. Το είπα και στην αρχή. Οι εργασίες για την ευημερία των ζώων θα πρέπει να επιταχυνθούν. Και με την θέσπιση κάποιων μέτρων και την επιλογή κάποιων λύσεων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την, τις πραγματικές δυνατότητες και το πόσο εφικτές είναι αυτές οι διατάξεις στην πράξη για τους γεωργούς. Να μην επιβάλλουμε υπερβολικά απαιτητικέ διατάξεις που θα είναι ανέφικτες στην πράξη. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε πολύ απαιτητικοί, μερικές φυσιολογικές διαδικασίες δεν επιδέχονται συντόμευσης. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι προσβλέπω σε αγαστή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια των νέων αρμοδιότητων που έχει και από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Θα ήθελα να έχουμε συχνές επαφές, όχι μόνο στην αρχή και στο τέλο τη Προεδρία για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων και για τον απολογισμό. Θα ήθελα να έχουμε τακτικέ επαφέ στο μέτρο που προχωρούν οι εργασίε στο Συμβούλιο, στο μέτρο που εξετάζουμε τι νομοθετικέ προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν όχι στην Ολομέλεια, τουλάχιστον ε, στα πλαίσια ε, αρχηγών πολιτικών ομάδων και προεδρίου θα μπορούσαμε να έχουμε επαφές για να εξετάσουμε τα πιο σημαντικά θέματα. Ή πριν από ένα Υπουργικό Συμβούλιο ή μετά για να ενημερωνόμαστε για την πορεία των εργασιών του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και να συντονιζόμαστε και δυνατόν να συμφωνούμε κιόλας. Σας ευχαριστώ. Uh, Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σας. Μα άρεσαν πολλά από αυτά τα οποία είπατε, γιατί πάνε στην κατεύθυνση που θέλουμε. Οπωσδήποτε η χρήση γης ε, μέσω της γεωργίας, ε, δασοκομείας και αλληλείας έχει μεγάλη σημασία στον 21ο αιώνα Πρέπει να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα οικοσυστήματα, το φυσικό κεφάλαιο και θα τα καταφέρουμε ή θα τα καταστρέψουμε. Αυτά είναι ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Είπατε πολλά πράγματα. Είναι πράγματι κρίμα πως η γεωργική πολιτική ε, αφορά κατά 90% τα λεφτά και όχι μια συνολική προσέγγιση το τι κάνει η Γεωργία για την κοινωνία και να αμυφθεί ακριβώς μια τέτοια επίδοση. Επίσης, να αναφερθήκατε ε, για το τι γίνεται ε, Παγκοσμίω, εμεί έχουμε ασχοληθεί με την εισαγωγή και την παράνομη εισαγωγή ξύλου από τους τις ε, τροπικές περιοχές και θα πρέπει να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα σύστημα. Ένα θέμα το οποίο αναφέρεται και πρέπει να μας απασχολήσει τα 30 εκατομμύρια εκτάρια τα οποία χρειαζόμαστε παγκοσμίω ε, για εισαγωγή ζωοτροφών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χρήση γης λοιπόν θα πρέπει να είναι ένα θέμα της ανθρωπότητας παγκόσμιο και στην επόμενη κλιματική διάσκεψη στην Νότια Αφρική. Αυτή η χρήση γης ε, θα είναι ένα σημαντικό θέμα. Και τα έμεσα αυτά αποτελέσματα επίσης πρέπει να συνυπολογιστούν, αλλιώς ε, δεν θα ε, προστατεύσουμε το κλίμα και δεν θα δούμε βεβαίω και την καταστροφή, την αλλαγή τερασίων εκτάσεων και τοπίων. Θα δεχτούμε την πρόσκλησή σας λοιπόν για επικοδομητική συνεργασία. Η Επιτροπή μας θέλει να σας βοηθήσει να έχετε μια επιτυχή προεδρία και είστε βεβαίως πάντα ευπρόσδεκτος εδώ πέρα. Αναφέρατε διάφορες διασκέψεις που θα οργανώσει η Προνική Προεδρία για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για σοκομεία και οπωσδήποτε θα έρθουν και διάφοροι ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς και την ομάδα σας και ευχόμαστε καλή επιτυχία τους ερχόμενους μήνες. Äh. λοιπόν, συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, το οποίο είναι ο προϋπολογισμός 2012. Και στην ώρα ήρθε και η Γιούτα Χάουγ, καλώς ήρθατε, η συγγήτρια, για να δούμε τι τρέχει εδώ στα δικά μας έχουμε περισσότερα λεφτά, λιγότερα λεφτά. Γιούτα, εσύ το είδες αυτό το θέμα, για πες μας. Ναι, ευχαριστώ. Ούτως ή άλλως, από αυτή την εβδομάδα υπάρχει το σχέδιο τοποθέτησης της Επιτροπής μας, μόνο στα αγγλικά, αλλά αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε πολύ σφιχτές προθεσμίες. Ξεκολουθούμε να μην έχουμε επίσημη απόφαση του Συμβουλίου, αλλά πρέπει να εργαστούμε με βάση μια τέτοια απόφαση. Υπάρχει μόνο μια απόφαση κορεπέρ που θα πρέπει μέχρι τις 25 Ιουλίου σε γραπτή διαδικασία να υπογραφεί από τους Υπουργούς και εμείς παριστάνουμε και θεωρούμε πως αυτό θα ήταν ε, το τέλος της πρώτης ανάγνωσης του Συμβουλίου. Τώρα, τι υπάρχει στο δικό μας το ψήφισμα. Εμείς λέμε ναι εντάξει, χαιρετίζουμε το ότι και το περιβάλλον και η δημόσια υγεία ανήκουν στη στρατηγική της Ευρώπης 2020, ούτως ή άλλως είμαστε υπέρ ε, μιας αηφόρου αποτελεσματικής οικονομίας, αλλά μετά αν δούμε τι έχει προτείνει η Κομισιόν από πλευράς ε, κονδυλίων στον προϋπολογισμό, βλέπουμε πως δεν πρόκειται καν για πάγωμα. Ονομαστικά, και τα έχω γράψει εγώ αυτά, μιλάμε για 2,6% αύξηση και 2,4% για τη δημόσια υγεία, αλλά γνωρίζουμε όλοι πως η Κομισιόν υπολογίζει έναν πληθωρισμό 2,9%. Αυτό σημαίνει, δηλαδή, εντάξει, είναι ένα πάγωμα ε, για να ακριβολογούμε κιόλα πρόκειται για μια μικρή μείωση. Και αυτό ισχύει και για τις υποχρεώσεις και για τις πληρωμές. Και αν δούμε μετά τι έχει κάνει το Συμβούλιο, με την πρόταση της Κομισιόν έχουμε και άλλη μείωση. Αλλά θα πω κάτι και για τις τροπολογίες. Αυτό το οποίο είναι σαφές είναι πως ήδη η Κομισιόν στο προσχέδιο ή μάλλον όχι, στο σχέ... όχι προσχέδιο, δεν υπάρχει πια, στο σχέδιο προϋπολογισμού, δημιουργεί τεχνητά περιθώρια μέσω του να μην δίνει τα assigned revenues στον ε, ΕΟΦ. Δηλαδή στο περιθώριο, στο 1α έχουμε ε, κάνα 2 εκατομμύρια παραπάνω εκεί που ανήκει ο ΕΟΦ. Ε, αυτό θα πρέπει να αναβελτιωθεί μετά. Αυτό το οποίο επίσης ε, γράφω εδώ πέρα και ούτως ή άλλως ε, εδώ και καιρό ισχύει αυτό, πώς θα πρέπει επιγόντως να έχουμε βελτίωση στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα κράτη-μέλη. Αλλά εντάξει, εμείς μπορούμε να κάνουμε όσο κήρυγμα θέμε, το ξέρουμε. Εάν δεν έχουμε αρκετό προσωπικό που θα ελέγχει την εφαρμογή, τότε δεν θα γίνει τίποτα. Και εκεί πέρα πράγματι ανησυχώ για το ότι η Κομισιόν Λόγω και αυτού του λαϊκισμού που λέει πρέπει να κόψουμε και γρήγορα άμεσα από τη διοίκηση, ε, υποτάσσεται σε αυτό και λέει ναι θέμε 5% λιγότερες θέσεις, θα αλλάξουμε το καταστατικό. Ε, εντάξει, το καταστατικό να αλλάξει. Αλλά μειώνετε μειώνεται όλο το κόστος του προσωπικού και εκεί πέρα έχω τις, ε, τις αμφιβολίες μου. Αν έχουμε συνολικά 5% λιγότερο προσωπικό, εκεί πέρα ξεκινάνε οι αμφιβολίες μου. Γιατί ξέρετε, δεν θα κόψουν ε, διευθυντές και γενικούς διευθυντές, θα κόψουν τους χαμηλόβαθμους, τους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά δηλαδή που θέμε. Και ελπίζω να έχουμε επαρκείς ε, πληροφορίες για να μπορέσουμε και εμείς να κινηθούμε αναλόγως. Ε, Μην γίνει δηλαδή αυτό. Το βλέπετε, αυτό δεν γίνεται μόνο στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και ΣΑΝΚΟ, αλλά και σε άλλες γενικές ε, διευθύνσεις. Και στην, και στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Τέλος πάντων τώρα αυτό δεν μας αφορά. Μας. Έχουμε δουλειές να κάνουμε, αλλά πρέπει να το έχουμε κατά νου και το έχω γράψει και στο ψήφισμα. Δεύτερον, το οποίο δεν ήταν δική μας αρμοδιότητα παλαιότερα, είναι τα τρόφιμα για τις μειονεκτικές ομάδες του πληθυσμού. Δεν είχαμε εδώ πέρα πότε πρόβλημα γιατί υπήρχαν πάντα αρκετά χρήματα στον προϋπολογισμό της Γεωργίας, αλλά μετά ένα κράτος μέλος, το οποίο το ξέρουμε εμείς οι δύο γιο, ποιο είναι, ε, κατήγγειλε αυτό το καθεστώς, δεν συμμετείχε ούτως ή άλλως ποτέ, δεν είχε πάρει ποτέ λεφτά από, αυτή, από αυτό το μέσο γιατί η Γερμανία δηλαδή είπε πως εμείς έχουμε κοινωνική πολιτική και ε, αυτό είναι δική μας δουλειά, είναι επικουρικότητα, δεν είναι θέμα αυτο το προϋπολογισμού, αλλά πολλά κράτη-μέλη εποφελήθηκαν από αυτό. Δεν ξέρω Ήρθε σε μένα η Κάριτας, διακονεί όλες οι κοινοφελείς οργανώσεις ε, που κάνουν αυτά τα συσίτια. Ε, ήρθαν και μου είπαν, μα κάντε κάτι, δεν είναι δυνατόν, ε, πρέπει να σπίσουμε να συμμετάσχει και η Γερμανία γιατί και εμείς δεν έχουμε λεφτά. Όμως η Γερμανία προσέφυγε στο δικαστήριο και το δικαστήριο είπε ναι, η Γερμανία έχει δίκιο πάμε πολύ πέρα από τη νομική βάση για την κοινή γεωργική πολιτική και άρα πρέπει να αλλάξει. Αλλά η Κομισιόν δεν έχει προτείνει άλλη νομική βάση, γι' αυτό προειδοποιούμε εδώ πέρα και πρέπει αυτό να γραφτεί στο 1α στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να πληρωθεί, αλλά με πολύ λιγότερα λεφτά. Και εκεί πέρα φοβάμαι, ειδικά σε αυτή την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε ούτως ή άλλως σε ολόκληρη την Ευρώπη, πως δεν θα υπάρχουν αρκετά λεφτά. Και πρέπει να παρακαλέσουμε την Κομισιόν εδώ πέρα, έτσι λίγο να κινηθεί κάπως γρήγορα για να έχουμε μια κανονική νομική βάση. Οπότε, επόμενο σημείο. Η καμπάνια HERB, ε, η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί δεν υπάρχει πλέον το Ταμείο Καπνού και παίρναμε τα λεφτά από τους καπνοκαλλιεργητές για να καταπολεμήσουμε την ε, κατανάλωση καπνού. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι είναι λογική αυτή η καμπάνια και με αυτά τα μέτρα ενημέρωσης Δεν μπορούμε να πούμε τώρα πως ε, έχουν ε, ενημερωθεί τόσο πολλοί οι νέοι για να μην ξεκινήσουν καν το κάπνισμα, το οποίο είναι το βασικότερο, για να το κόψουν. Εν πάση περιπτώσει, τώρα υπάρχει το πρόγραμμα δράσης για την υγεία και, και από εκεί πέρα θα χρηματοδοτηθεί εκστρατεία κατά του καπνίσματος, ε, για τα, από θα λάβουμε 10 εκατομμύρια Επίσης συζητάμε από την Κομισιόν επιτέλους να υποβάλει το τροποποιημένο φύλλο προϋπολογισμού για την φαρμακοεπαγρύπνηση, γιατί ξέρουμε πως ο ΕΟΦ, ο Ευρωπαϊκός, θα έχει περισσότερες αποστολές και θέλει περισσότερο προσωπικό, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν έχουμε αυτό το φύλλο το οικονομικό, γιατί πρέπει να περιγράφεται πόσο προσωπικό χρειάζονται και λεφτά. η υπηρεσία εξωτερική δράσης και ΕΚΑ και εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα με το προσωπικό. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα. Απευθύνω πάλι προειδοποίηση στην Κομισιόν. Τώρα, στην προθεσμία που έχουμε εμείς για τροπολογίες που είναι αύριο και για το σχέδιο ψηφίσματος και για και στον ίδιο τον προϋπολογισμό, δεν έχω κάνει τίποτα όσον αφορά το ύψος των τελών της ΕΦΣΑ. Πριν από δύο χρόνια είχαμε πει, είχαμε προειδοποιήσει πως πρέπει κάτι να γίνει και αναγκάσαμε την Κομισιόν και μας ε, έστειλε μία μελέτη για τις ε, πιθανότητες ε, τελών της ΕΦΣΑ και εκεί πέρα μείναν τα πράγματα. Έγινε μία συζήτηση στην Επιτροπή, όλες οι ομάδες ήταν θετικές για αυτό το ύψος των τελών που δεν θα χρηματοδοτούσαν βεβαίως Πλήρω την ΕΦΣΑ, αλλά τουλάχιστον τα πράγματα τα οποία κάνει για την βιομηχανία τουλάχιστον η ΕΦΣΑ. Αυτά να τα πληρώνει η βιομηχανία. Τώρα τα χρειαζόμαστε αυτά τα τέλη, γιατί ξέρετε, χρειαζόμαστε την πρόταση για να ακολουθεί η κανονική νομοθετική διαδικασία και... Θα ήθελα τώρα να ξέρω, είναι ε, διατεθειμένη η Κομισιόν ε, να μας τα στείλει εγκαίρως. Αλλιώς πάλι θα ε, πάνε στο αποθεματικό της ανάλογης γενικής διεύθυνσης. Μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου πρέπει να γίνει αυτό. Ε, απλά το αναφέρω ξανά εδώ μέσα. Τροπολογίες που υπέβαλα εγώ. Όπως είπα μπορούν όλοι να υποβάλουν τροπολογίες η προθεσμία είναι μέχρι τις 15 Εβδόμου. Για τον ΕΟΦ λοιπόν, ξανά αυτά τα καθορισμένα έσοδα στο σχέδιο προεπιλογισμού της ΕΜΑ. Μετά για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Έχουμε ξανά το σχέδιο προπολογισμού, τα λεφτά δηλαδή που πάλι έκοψε το Συμβούλιο και διέγραψε και θέσεις του προπολογισμού τις οποίες εμείς ε, επανεισάγαμε. Για την ΕΦΣΑ λοιπόν και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών και την ΕΚΑ Ευρωπαϊκή Χημική Υπηρεσία, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών Ουσιών. Έχουμε το σχέδιο προϋπολογισμού και για πρώτη φορά και παραβιάζω μία αρχή μου αλλά θεωρώ πως πρέπει να γίνει εδώ πέρα γιατί η Κομισιόν κάθε φορά είναι σκληρή και ε, δεν υποχωρεί η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού. Για πρώτη φορά θα καταθέσουμε τροπολογία για το οργανόγραμμα και εκεί πέρα τις 10 θέσεις που χρειάζεται η ΕΚΑ έχουμε προσθέσει. Η Κομισιόν δεν θέλει αυτές τις ε, θέσεις για το Συμβούλιο εννοείται καθόλου. Αλλά ούτως ή άλλως δεν επηρεάζουν τον προϋπολογισμό γιατί θα πληρωθούν από τα τέλη. Το θέμα είναι οι νέες αποστολές που έχει η αίμα να μπορεί να ε, τις καλύψει κιόλας και δεν γίνεται αλλιώ. Γιατί ξέρετε, είναι θέματα τα οποία Πρέπει να κάνει λοιπόν αυτές τις επιστημονικές αξιολογίες. Αλλά αυτά τα πληρώνουν οι επιχειρήσεις μέσω των τελών. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να μην ε, δημιουργηθούν αυτές οι δέκα θέσεις. Τις Βάλαμε λοιπόν εμείς τώρα, αν μπορεί να θυμηθεί κανείς την τελευταία διαδικασία του προπολογισμού που έλεγα εγώ όχι, πρέπει να παραδεχτούμε πως η Κομισιόν έχει τη γενική εποπτεία, πως μπορεί να κάνει περισσότερα και θα έρθει μετά με έναν διορθωτικό προϋπολογισμό. Τώρα πρέπει να παραβώ αυτή την αρχή μου. Οπότε θα δημιουργήσουμε αυτές τις 9-10 νέες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών Ουσιών και όπως σας είπα δεν κοστίζει τίποτα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, δεν χρειαζόμαστε κανένα περιθώριο, δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Τις τροπολογίες τώρα δεν θα τις αναφέρω όλες, το θέμα είναι απλά για να απορρίψουμε τις περικοπές που θέλει το Συμβούλιο για να παραμείνουμε τουλάχιστον στην πρόταση της Κομισιόν. Τίποτα άλλο δεν έχω αλλάξει. Οπότε θα επανέλθουμε στην πρόταση της ε, Κομισιόν ε, για τον ΕΟΦ. Και ο ΕΟΦ έχει τα δικά του καθορισμένα έσοδα. Πριν τελειώσω να πω ακόμα πως ο Τόμας Ούλμερ ε, μου έγραψε και μου είπε πως ε, θα απουσιάζει σήμερα, αλλά υποστηρίζει αυτά τα οποία έχω γράψει στο ψήφισμα και πιθανώς το ΕΛΚ δεν θα καταθέσει τροπολογίες ε, για το ψήφισμα και είμαι πολύ ικανοποιημένη αλλά θα ακούσουμε και τις απαντήσεις κομισιών. Αυτά ήθελα εγώ να πω. Τώρα πήρ κατά βούληση. Ευχαριστούμε Γιούτα. Βασιζόμαστε στη δική σου την πείρα και την τεχνογνωσία. Produkt, äh, was nennt, wir wissen ε, χωρίς λεφτά δεν γίνεται τίποτα. Οπότε είναι σημαντικός ο προπολογισμό. Äh, και δεν ξέρω καθένας βεβαίως πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό και οι αδυναμίες του κοινοτικού προπολογισμού. Κυρίως σε ευχαριστούμε για τις πέντε υπηρεσίες που έχουμε εμείς, που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έχουμε παρατηρήσει πόσο ευγνώμονες είναι στο Λονδίνο, στην Πάρμα, στο Ελσίνκι. Γιατί ε, ξέρετε πως δεν είναι τα αγαπημένα παιδιά του Συμβουλίου. Δεν τους ε, αρέσουν εκεί στο Συμβούλιο. Και το Κοινοβούλιο πρέπει ως δημοσιονομική αρχή να διατηρεί και να γνωρίζει τις ανάγκες αυτών των υπηρεσιών. Λες πως πρέπει να τις βοηθήσουμε όλες αυτές και πρέπει να μπορούμε και να το κάνουμε. Κάποιοι, κάποια από αυτά έχουν έσοδα και αναφέρθηκε και το μέγεθος των εσόδων και καλό είναι να υπάρχει μια σαφήνεια πόση αυτοχρηματοδότηση ε, υπάρχει για να μην ε, κρέμονται συνέχεια από τον προπολογισμό και τον φορολογούμενο. Για το γενικό προϋπολογισμό είπες πως αν είμαστε ευγενικοί είναι στάσιμος, ε, ε, αν το δούμε προσεκτικά μειώνεται. Το είπανε και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αυτό. Χτες το έστειλα αυτό το οποίο ε, μου έστειλε στα μέλη της Επιτροπής, γιατί η Κομισιόν λέει συνολικά ο προπολογισμό γίνεται πρασινότερος, αλλά ε, αυτό ήταν βεβαίως ε, οι μεσοπρόθεσμες ε, δημοσιονομικές προοπτικές, όχι το 2012. Και δεν γίνεται, νομίζω, πολύ πιο πράσινος, αλλά... Εδώ πέρα βλέπουμε στο 2012, μιλάμε για μικρά ποσά και η εκτίμησή σου ήταν πως είναι και μείον και όχι συν. Οπότε θα δούμε τις τροπολογίες σου. Πράγματι αύριο είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες και 8 Σεπτεμβρίου έχουμε μια επιπλέον συνεδρίαση με την Επιτροπή Προϋπολογισμού Τώρα ο κ. Κεπράντη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τη Γιούτα Χάουκα για όλη τη δουλειά που έκανε Σύμφωνα με τα περισσότερα από τα συμπεράσματά σα, ε, Πρόεδρε, για το Γενικό Προπολογισμό, Νομίζω ότι έχει δίκιο η Κομισιόν ότι το περισσότερο από το περσίνισμα θα γίνει στους άλλους τομείς, αλλά εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε επαρκεί πόρους ε, στους συγκεκριμένε γραμμές προπολογισμού. Κάτι που θέλω να τονίσω είναι η σημασία της, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Ε, θα αναλάβει νέα καθήκοντα αυτός ο οργανισμός. Και είναι γνωστό ότι είναι ένα από, το, από τους καλύτερους οργανισμούς ε, ως προς την ε, διαχείρισή του, προς τη δίκησή του που έχουμε στην Ευρώπη και σήμερα πάλι βρίσκεται αντιμέτωπος με περικοπές και έχουμε πολύ μικρά ποσά για αυτά τα επιπλέον καθήκοντα Χτες ε, ήρθε και το Υπουργό ε, περιβαλλοντό, πάλι μα τόνισε πως σημαντικά είναι τα νέα δεδομένα, τα νέα στοιχεία και πάλι εξαρτόμαστε από τον οργανισμό μα ε, στην Κοπενχάγη για τη συλλογή αυτών των στοιχείων. Θέλω να τονίσω λοιπόν το πόσο σημαντικό είναι και ελπίζω εμεί από τη Σκοπιά του Κοινοβουλίου να μπορούμε να διασφαλίσουμε αυτού τους πρόσθετου πόρου για αυτό το πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό οργανισμό. Ευχαριστώ. ευχαριστώ τη Γιούτα. Ζητάμε ε, προσωπικό γιατί μας λένε τα ΜΜΕ πως ε, υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίοι υπάλληλοι. Και το θέμα λοιπόν είναι πόσο είναι το προσωπικό για τον έλεγχο ε, της νομοθεσίας αυτής. Γιατί αν μπορούμε να απαντήσουμε πως αυτοί είναι οι άνθρωποι που ελέγχουν αυτά τα πράγματα, θα είναι σαφές νομίζω, θα μπορούμε να απαντήσουμε κάτι. Δηλαδή τη στιγμή που μπορώ να πω πως ο αυστριακός προϋπολογισμός κατέτος ε, έχει το ύψος ε, του ευρωπαϊκού, ε, σταματάει ο κόσμος. Γιατί συνήθως ακούνε κάτι τερατοδίες από πλευράς αριθμών. Μάλιστα. Έχω ένα ερώτημα γιατί χτύπησαν τα καμπανάκια κατά τη διάρκεια της χρονιάς για την ε, προστασία του κλίματος, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και διεθνείς υποχρεώσεις. για την προστασία του κλίματος, για τη βιοπικιλότητα. Είναι σίγουρο πως ε, θα πληρώσουμε ε, αυτές τις υποχρεώσεις. Γιούτα, πριν ε, ξαναμιλήσεις, καλό είναι να ακούσουμε την Κομισιόν. Έχουμε εδώ λοιπόν την Αν Μποεγιό. Ναι. Όχι. Ναι. Εκπληξούλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προέρχομαι από τη ΓΑΜΑ Περιβάλλοντος. Θα αναφερθώ σε ορισμένα από τα θέματα τα οποία τέθηκαν σε ό,τι αφορά την πρόταση της Κομισιόν υπό το σχέδιο προπολογισμού. Ο προπολογισμό για το περιβάλλον και για την κλιματική δράση υπό το τίτλο 7 αυξάνεται κατά 2,6%. Αλλά θέλω να τονίσω και το ότι οι περισσότερε από αυτέ τι δαπάνε είναι υπό το πρόγραμμα LIFE και η Κομισιόν έχει προτείνει αύξηση 4,3% για το πρόγραμμα αυτό. Αυτό είναι πάνω από το 2% λοιπόν συνολικά. Και σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, η πρόταση της Κομισιόν για το σχέδιο προϋπολογισμού περιλαμβάνει προτάσεις ε, για επιπλέον προσωπικό, για την επιτέλεση νέων καθηκόντων, συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα και για το κλίμα. Τώρα για την εφαρμογή της νομοθεσίας ε, και του αριθμού του προσωπικού. Μπορούμε να δώσουμε τα αριθμητικά στοιχεία των ανταμών που εργάζονται στη ΓΑΜΑ περιβάλλοντος. Ε, είναι σε μια συγκεκριμένη ε, διεύθυνση, δεν είναι δύσκολο να βρούμε αυτά τα στοιχεία και καλωσορίζω την έκκληση που υπάρχει στο ψήφισμα απέναντι στα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί και αυτά είναι προτεραιότητα για την Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Thank you. Yeah, Χιούτα. Ε, ε, απαντήθηκαν τα περισσότερα. Γίνεται πιο πράσινος ο προϋπολογισμός. Αυτό είναι το σχέδιο για το... τις πολιετής προοπτικές. Αλλά πρέπει να δούμε την νομοθεσία και μπορώ από τώρα να ζητήσω το εξής από τους συναδέλφους. Όταν μιλάμε για τη γεωργία, όταν μιλάμε για την νομοθεσία την περιφερειακή, πρέπει να φροντίσουμε να μείνουν όλα αυτά μέσα. Ε, ήδη ακούμε τις διαμαρτυρίες απ' έξω. Στον πρώτο πυλώνα το 30% αυτό το πρασίνισμα. Δεν θα γίνει λένε αποδεκτό. Εκεί πρέπει να πιάσουμε τους συναδέλφους στην Επιτροπή Γεωργίας και να τους πούμε όχι θα το κάνετε. Τα είχαμε συζητήσει όλα αυτά ως κοινοβούλιο με την έκθεση ΣΟΥΡ, αλλά πρέπει να γίνουν και νόμος. έστω και αν ο Επίτροπος μετά, ο κύριος Χάν κάνει τις ε, προτάσεις του για την περιφερειακή πολιτική, εντάξει, να τις δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει με τις επιβλαβείς επιδοτήσεις. Λοεκθέσεις γράφουμε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και τα νούμερα. θα ζητήσουμε τις Γενικές Διευθύνσεις ε, να κάνουν κάτι τέτοιο για μας, για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, να ξέρουμε πόσο επιβλαβής ε, είναι, ε, ποιες είναι οι επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις. Αυτά, αυτά για το μέλλον, όπως είπα. Και στον τωρινό προϋπολογισμό για τις διεθνείς υποχρεώσεις υπάρχουν περισσότερα από ό,τι στον προηγούμενο και και είναι πάντα το ερώτημα πώς μαζεύει η Κομισιόν αυτά τα οποία υποσχέθηκαν τα κράτη-μέλη. Το έχουμε ζητήσει παραπάνω από μία φορές. Θέμε στοιχεία. Ποιος πλήρωσε, ποιος δεν πλήρωσε, ε, για να κάνουμε και κάτι. Ε, στη χώρα μας. Δεν ξέρω τι έγινε με τη Γερμανία. Αλλά δεν, δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Αυτή είναι η δυσκολία. Τέλο πάντων, δεν ξέρω ποιο τα είδε. Για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο τα έχουν εκτός του συνολικού πλαισίου εκεί και λένε χωρίς νούμερα, χωρίς μεμονωμένα νούμερα. Και αυτό είναι όμως άρα οι ε, υποσχέσεις αυτού του μέσου που πρέπει να εκταμιευθούν από τα κράτη-μέλη. Δεν το έχω δει το, το μέσο ακόμα, αλλά πρέπει, να ασχοληθούμε με αυτό. Αλλά όπως σας είπα όλα αυτά είναι για το, για το 12 ε, και δεν έχουν ετοιμαστεί ακόμα, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, ναι, είναι ξεχωριστή κάστα αυτοί που ασχολούνται με τον προπολογισμό όχι πολύ αγαπητή, αλλά παρόλα αυτά απαραίτητη. Έχεις και το μονοπόλιο εδώ στην Επιτροπή, γιατί, ξέρεις, είναι σημαντικό να κοιτάει κανείς ε, ακριβώς ε, τον προπολογισμό. Εμείς αποφασίζουμε πολιτικές και ιδέες, αλλά η υλοποίηση μετά είναι άλλη. Ωραία. Λοιπόν, Ελπίζω. Να έχουμε μια βοήθεια, μια συνεισφορά. Εκτός από το συνάδελφο που προσφέρθηκε, εσύ φοβούμαι ότι θα τα επομιστείς όλα. Ωραία. Οπότε ευχαριστούμε Γιούτα και συνεχίζουμε παρακάτω, σημείο 19. Υποβολή της ενδιάμεσης αναθεώρησης του κανονισμού LIFE. Ο Τίμο Μάκελα είναι εδώ. Γενικός Διευθυντής ε, Διεθνών Σχέσεων του προγράμματος Live στη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ που δίνετε την ευκαιρία αυτή στην Κομισιόν να σας παρουσιάσει εν συντομία το πρόγραμμα LIFE, την ενδιάμεση αναθεώρηση του προγράμματος 2007-2009 η οποία ολοκληρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν λίγους μήνες και παρουσιάζεται τώρα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αυτή η αναθεώρηση βασίζεται στην ε, πρόσληψη ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων για να γίνει αναθεώρηση για την Κομισιόν ε, βάσει συμμετοχής ε, πολλών ενδιαφερομένων μερών, διαβούλευσης με πολλά ενδιαφερόμενα μέρη. Ε, το κύριο συμπέρασμα της ενδιάμεσης αναθεώρησης είναι ότι το πρόγραμμα LIFE ήταν ένα πολύ επιτυχές μέσο από τη στιγμή που σχεδιάστηκε, από τη στιγμή που ξεκίνησε, το 1992. Πάνω από 3.000 προγράμματα χρηματοδοτήθηκαν υπό το LIFE και συνείσφεραν με επιτυχία στο να καλυφθούν οι ανάγκες της περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το κύριο πόρισμα της ε, ενδιάμεσης αξιολόγηση. Τώρα, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο γιατί. Γιατί θεώρησαν οι ότι το LIFE ε, είναι ένα επιτυχές εργαλείο. Καταρχήν, διαδραμάτισε ένα σημαντικό ρόλο στην δημιουργία και στην ε, εφαρμογή της Οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οικοσυστήματα και για την προστασία των πτηνών και των σχετικών δικτύων. Επίσης, υπήρξε ένα πραγματικό εργαστήριο για την εφαρμογή νέων προσεγγίσεων για να προωθήσουμε την εφαρμογή των πλέον απαιτητικών νομοθετημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η οδηγία πλαισίου για το νερό. Και τρίτον, αύξησε, σύμφωνα με την αξιολόγηση, την ευαισθητοποίηση των πολιτών για περιβαλλοντικά θέματα και την πρόσβασή τους σε περιβαλλοντικές πληροφορίες. Για πολλούς, το live είναι το μόνο μέσο που αφιερώνεται αποκλειστικά στο περιβάλλον που αφορά αποκλειστικά το περιβάλλον και πραγματικά αποτελεί σημείο αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τι περιβαλλοντικέ δαπάνε. Φυσικά η διάμεση αναθεώρηση Εντοπίζει επίσης τομείς όπου θα μπορούσε να βελτιωθεί το πρόγραμμα. Παραδείγματος χάρη. Προτείνεται μια καλύτερη εστίαση και καλύτερη ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Κάτι τέτοιο θα βοηθούσε στο να έχει καλύτερο αντίκτυπο το πρόγραμμα, κυρίω σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική πολιτική και την ε, διαχείριση. Η διακυβέρνηση, αν Δεύτερον, συμπεραίνεται ότι ορισμένα σκέλη του προγράμματος θα μπορούσαν να προσδιοριστούν ε, καλύτερα για να είναι πιο επιτυχή. Παραδείγματο χάρη, ε, το σκελός για τη βιοποικιλότητα του live θα μπορούσε να επικεντρωθεί περισσότερο στην επίδειξη καλύτερων πρακτικών. για να είναι πιο αποτελεσματικό. Και επίσης ε, υπάρχει και το συμπέρασμα ότι το σκέλος ε, ενημέρωσης και επικοινωνίας ε, του live, που είναι ένα νέο σκέλος στο σημερινό πρόγραμμα, δεν έχει κατανοηθεί πλήρως και ούτε έχει χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης, οικοδόμηση συνεργειών με άλλα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν κάτι αρκετά δύσκολο και υπήρξαν ε, όρια στην επέκταση των ε, προγραμμάτων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, ορισμένα από αυτά τα χωρίσματα και συγκεκριμένα οι ελλείψεις ήδη λαμβάνονται υπόψη ε, κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος υπό αυτές τις δημοσιονομικές προοπτικές, αλλά φυσικά Τώρα σχεδιάζουμε και τον πιθανό διάδοχο του live. Αν μου, επιτρέψετε, αν μου επιτρέπετε, mm. θέλω να αναφερθώ και στο έργο της Κομισιόν για τις μελλοντικέ δημοσιονομικές προοπτικές. Βάσει της ανακοίνωσης της Κομισιόν ε, για τον προπολογισμό για την Ευρώπη του 2020, απόφαση που ελήφθη από την Κομισιόν στις 20 Ιουνίου. Στην ανακοίνωση αυτή η Κομισιόν προτείνει ένα μέσο που θα διαδεχτεί το live με ένα προπολογισμό 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάτι τέτοιο αποτελεί αύξηση του σημερινού επίπεδου προπολογισμού και σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν θα διαιρεθεί αυτό το ποσό μεταξύ του περιβαλλοντικού σκέλους 2,4 ε, και το υπόλοιπο 1,8 για την κλιματική αλλαγή. Η Κομισιόν πιστεύει ότι πρέπει να παραμείνει η στις περιβαλλοντικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κλιματική αλλαγή, βιοπικιλότητα, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα των πόρων και πρασίνισμα των οικονομιών μας συνολικά και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν θεωρεί ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς αηφόρο, διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος. Και αυτό συνάδει με τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπης 2020. Υπό το νέο μέσο, η Κομισιόν, πέρα από την περιοδοσιακή προσέγγιση, πέρα από το περιοδοσιακό project, ε, σχεδιάζει και ένα νέο project που θα συμπεριληφθεί στο LIFE, το οποίο αποκαλείται Integrated Project, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ο στόχος θα είναι να προωθηθούν ορισμένα από τα προγράμματα και να προέρθουν ε, να προωθεί χρηματοδότηση και άλλες πηγές ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από περιοχές ε, των κρατών μελών για να δεθούν σε εφαρμογή οι πολιτικές τη Ευρωπαϊκής Ένωση για το περιβάλλον, παραδείγματο χάρη για την βιοπικιλότητα, το είδωρ και για τα απόβλητα. Η μελέτη δικτύπου τη πρόταση αυτή είναι υπό ολοκλήρωση για να μπορέσουμε στη συνέχεια να παρουσιάσουμε μια πιο συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση του μέσου που θα ακολουθήσει το LIFE αναμένεται περί τα τέλη του έτους, Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Για να ολοκληρώσω. Το live, σύμφωνα με αυτή την ενδιάμεση αναθεώρηση, ήταν και θα είναι στο μέλλον, στο μέλλον με συγχωρείτε, ένα χρήσιμο και σημαντικό μέσο για την προώθηση της ανάπτυξης και της εφαρμογής των περιβαλλοντικών πολιτικών της Ένωσης και για την επιδείξη των βέλτιστων πρακτικών. Σας ευχαριστώ. Σα danke, Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε για την συνοπτική υποβολή της ενδιάμεσης αναθεώρησης του κανονισμού LIFE, που είναι το μοναδικό όργανο τέτοιου είδους που έχουμε για την περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης. Και σίγουρα φαίνεται από την ενδιάμεση αναθεώρηση ότι ο κανονισμός αυτός ε, έχει τύχει πολύ επιτυχημένης εφαρμογής. Φαντάζομαι θα υπάρχει και ένα πρόγραμμα παρακολούθησης, 3,2 δις, που θα κατανεμηθεί θα κατανεμηθούν σε μέτρα, ειδικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά όπως είδαμε θα πρέπει και άλλες δημοσιονομικές γραμμές ε, να τροφοδοτήσουν το live γιατί έχει αυξημένες ανάγκες. Υπάρχουν παρατηρήσεις ή ερωτήσεις ε, προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μια και θα προβείτε στην ενδιάμεση αναθεώρηση για το έκτο περιβαλλοντικό πρόγραμμα για το περιβάλλον, θα ήθελα να σας ρωτήσω, σκοπεύετε να υποβάλλετε αυτή την αναθεώρηση πριν το καλοκαίρι ή θα περιμένετε το φθινόπωρο για το έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, την αξιολόγηση επιπτώσεων για το έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Πότε σκοπεύετε να μας το υποβάλλετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώνει αυτή τη στιγμή την αξιολόγηση του έκτου περιβαλλοντικού προγράμματος δράσης, που είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα και μια και έχουμε ήδη φτάσει στα μέσα Ιουλίου, μάλλον αδύνατο να υποβληθεί η αξιολόγηση πριν τις θερινές διακοπές. Κατά πάσα πιθανότητα μέσως μετά την επιστροφή από τις θερινές διακοπές θα είναι έτοιμο. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, έχει περάσει από τις εσωτερικές διαβουλεύσεις. Δεν θέλω να δεσμεύσω τους συναδέλφους, πάντως φαντάζομαι ότι λίγες εβδομάδες μετά τις θερινές διακοπές θα μπορέσουμε να το υποβάλουμε. Καλώς. Αν δεν κάνω λάθος, η Πολωνική Προεδρία θα ασχοληθεί με την αξιολόγηση, οπότε θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια και ενέργειες, μεγάλη ενέργεια. Ελπίζω αμέσως μετά το καλοκαίρι να είναι έτοιμο για να υποβληθεί στο Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις προς τον κύριο Μακελάιναν. Γι' αυτό μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο, αλλά ίσως ε, ε, προχωράμε με ταχύς ρυθμούς και δεν είναι ακόμη εκπρόσωπος επιτροπής ή όχι. Όχι, εντάξει. Προχωρούμε στο σημείο 20. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον Γενικό Διευθυντή που είναι εκεί ο πρόσωπος στην Επιτροπή μας. Την τελευταία φορά που μας κάνατε παρουσίαση η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Είχαμε μια πολύ πρωτότυπη ιδέα να, να συναντηθούμε εκτός Βρυξελών και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η εμπειρία και η διάσκεψη εκείνη. Έτσι δεν είναι Ρίτσα Ζέμπερ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνάντηση. Και μία από τις ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν τι γίνεται όταν ένας βουλευτής κάνει μια ερώτηση και μετά φεύγει και δεν είναι παρόν στην απάντηση. Δύσκολο. Δύσκολο ερώτημα. Βέβαια, παρόλο που δεν έχουμε πολλούς βουλευτές, η βοηθή τους είναι εδώ, οπότε δεν θα πάει τίποτα χαμένο. Είναι η τελευταία συνεδρία της Επιτροπής μας πριν τις θερινές διακοπές, γι' αυτό και είναι κάπως αραιό κατοικημένη η αίθουσα. Παρ' όλα αυτά, θα ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον την τρίτη έκθεση παρακολούθησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά την ανακοίνωση για τη λειψιδρία και την ξηρασία στην Ευρώπη. Γιατί η λειψιδρία και η ξηρασία προβληματίζουν πολύ σοβαρά τις χώρες και τις περιφέρειες και οι συνέπειές τους είναι μερικές φορές ολέθριες. Ο κύριος Φάλκεμπερκ θα μας υποβάλει την έκθεση και θα δούμε μετά τις απαντήσεις. Ευχαριστώ. Είναι αλήθεια ότι την τελευταία φορά που παρευρισκόμουν εδώ ήταν ε, πλήρης η αίθουσα. Είχε πολύ περισσότερο κόσμο από τη σήμερα. Πάντως, ε, εν ώψη τη συζήτηση για το είδωρ, ε, όπω είπατε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Τώρα, εισαγωγικά, θα σας μιλήσω εν συντομία για την τρίτη έκθεση αλλά θα δράξω την ευκαιρία να σας πω και πώς σκοπεύουμε να προωθήσουμε το θέμα του ύδατος. Η τρίτη έκθεση που έχετε ενωπιόν σας, ουσιαστικά τι μας λέει. Ότι η κατάσταση επιδεινώνεται, αυξάνονται οι ανησυχίες, βλέπουμε ότι δεν έχουμε λειψιδρία μόνο στην Νότια Ευρώπη, αλλά είναι και κάτι κοινό, είναι ένα κοινό φαινομένο πάνω κάτω σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης. Με εξαίρεση κάποιων ε, περιοχών ε, στο βορρά της Ένωσης, ε, όπου έχουμε και μικρότερο πληθυσμό. Έχουμε χώρες, Τσεχία, Κύπρο, Προμάλτα να μας αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν συνεχή ζητήματα, σοβαρά ζητήματα λειψιδρίας και περισσότερα κράτη-μέλη τώρα αναφέρουν ότι έχουν ξηρασία και επίπεδα βροχοπτώσεων χαμηλότερα από ότι ο μακροπρόθεσμος όρος Γαλλία, Ουγγαρία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε ευρία γκάμα χωρών και περιλαμβάνονται και ορισμένα από τα μεγάλα κράτη-μέλη. Και ε, Βέλγιο, κάτω χώρες και Ηνωμένο Βασίλειο. Ότι έχουν ε, καταγράψει τις χειρότερες ξηρασίες ε, σε σχέση με τα τελευταία έτη. Έτσι λοιπόν ε, το θέμα του νερού παραμένει ενσχετικό στην Ευρώπη. Αλλά βέβαια αν δούμε την ευρύτερη εικόνα παγκοσμίω, συνειδητοποιούμε ότι έχουμε δισεκατομμύρια σε αυτό τον πλανήτη σήμερα που σε καθημερινή βάση δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο και ποιοτικό νερό και μπορείτε να φανταστείτε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε στην εκθεσή μας ότι δεν πρόκειται απλώς για περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά ότι το θέμα αυτό έχει και οικονομικές επιπτώσεις σε τομείς όπως η γεωργία, ο τουρισμός, στο, η βιομηχανία, για την ενέργεια και για τις μεταφορές. Και εν τέλει θα θίξει και την ανταγωνιστικότητα και την εσωτερική αγορά. Σημειώνουμε στην έκθεση ότι αρκετά κρατημέλη έχουν λάβει μέτρα, κάποια κρατημέλη έχουν λάβει μέτρα. Υποστηρίζουμε το βασικό προσανατολισμό να εργαστούμε για μέτρα που αφορούν τη ζήτηση, δηλαδή να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιούμε πιο αποτελεσματικά το νερό, πριν ε, να αρχίσουμε να εργαζόμαστε για νέα με νερό όπως είναι μεταφορές, η αφαλάτωση, γιατί πιστεύουμε ότι και τα δύο αυτά θα έχουν ε, και άλλες επιπτώσεις, ε, πρόσθετες επιπτώσεις για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και θα επιφέρουν και περαιτέρω περιβαλλοντικά προβλήματα. Τώρα, τι θέλουμε και τι σκοπεύουμε να κάνουμε αρχίσαμε να εργαζόμαστε για ένα ευρωπαϊκό blueprint ε, για το είδωρ. Θα έχουμε τον πίνακα Συμβουλίου και Κοινοβουλίου μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους ε, και εργαζόμαστε για αυτή την ε, συνολική προσέγγιση για θέματα ύδατος. Και βασικά χρησιμοποιούμε τέσσερα είδη ανάλυσης, ε, δηλαδή ε, βλέπουμε πώς γίνεται η διαχείριση, πώς, ποια είναι τα σχέδια διαχείρισης των ε, λεκάνων απορροής των ποταμών, θα έπρεπε να συμμετέχουν τα κρατημέλη, αλλά δυστυχώς έχουμε τέσσερα-πέντε κρατημέλη που δεν μας έχουν στείλει αυτά τα σχέδια για τη διαχείριση των λεκανών προϊόντων ποταμών εμά στην Κομισιόν. Δεύτερη αξιολόγηση που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι ένας έλεγχος ε, καταλληλότητας ε, για την πολιτική του νερού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχετική νομοθεσία, να δούμε αν ε, υπάρχει νομοθεσία στα κράτη-μέλη και να δούμε τι μπορεί να γίνει διαφορετικά, όπου χρειαστεί να υπάρχει streamlining και συμπλήρωση της νομοθεσίας. Επίσης, εξετάζουμε ε, την έκθεση για την πολιτική, για τη λειψιδρία και την ξηρασία και εξετάζουμε το πόσο ευάλωτη είναι η υδάτινη πόρη στην κλιματική αλλαγή. Γιατί γνωρίζουμε φυσικά ότι και η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε προσθέτη πίεση. Τώρα, να σας πω δύο λόγια σε σχέση με το blueprint και τι θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν με το σχέδιο αυτό να αξιολογήσουμε όλους τους τομείς ε, που έθιξα, αλλά υπάρχουν 7 τομείς που θα περιλαμβάνονται σε αυτό το blueprint, σε αυτό το σχέδιο. Θα πρέπει να δούμε τη διαχείριση των γεών. Ίσως ε, να σας εκπλήσει ότι το πρώτο σημείο που αναφέρω όταν μιλώ για το νερό είναι η γη, αλλά πιστεύουμε ότι για να έχουμε μια πολιτική για το είδωρο είναι σημαντικό να εξετάσουμε θέμα όπως ε, η διαχείριση του εδάφους, ε, βιώσιμα στήματα αποχέτευσης, ε, η αναδάσωση και τι όλα αυτά θα θίξουν την διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων, τη διαθεσιμότητα του νερού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαχείριση λοιπόν των γεών και τα θέματα που σας ανέφερα θα είναι η προ... ο πρώτος μεγάλος τομέας που θα πρέπει να αναλύσουμε. Δεύτερον, όπως ε, πάντα, όπως σε κάθε περίπτωση που έχουμε λειψιδρία, θα πρέπει να έχουμε μηχανισμούς στην αγορά και ο καλύτερος μηχανισμός στην αγορά που έχουμε είναι η τιμή. Θα πρέπει να εργαστούμε λοιπόν σε θέματα τιμολόγησης, να εσωτερικοποιήσουμε το κόστος ε, της χρήσης του νερού, θα πρέπει να δούμε το θέμα της ε, μόλυνσης του νερού. Είναι επίσης ε, καλό το ότι βλέπουμε στη σημερινή έκθεση ότι όλο και περισσότερα κράτη-μέλη συμπεριλαμβάνουν πολιτικές τιμολόγησης για το νερό. Το νερό δεν ε, είναι πλέον ένα δωρεάν αγαθό που μπορεί να βγάλει απλώς κανείς από ένα πηγάδι και να το χρησιμοποιήσει όπως θέλει, κατά βούληση και χωρίς κόστος. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η χρήση του νερού έχει κόστος και το κόστος αυτό πρέπει να αντικατοπτρίσει αν θέλουμε να είμαστε πιο αποδοτικοί. Έτσι, λοιπόν, θα συνεχίσουμε να συζητούμε την ανάγκη για τιμολόγηση, επιβολή φόρων, την εξάλληψη των επιβλαβών ε, ουσιών και επίσης να υπάρξουν ε, και συστήματα κατανομής νερού στην Ευρώπη όπου έχουμε ιδιαίτερα ε, έντονα φαινόμενα λειψιδρίας. Επίσης θα πρέπει να δούμε την ε, αποδοτικότητα του ύδατος και προκειμένου να αναπτύξουμε αυτή την αποδοτικότητα ελπίζουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τους λογαριασμούς οικοσυστήματος και υδατός θα πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τους διάφορους ε, τομείς, τις διάφορες περιοχές, με συγχωρείτε, στην Ευρώπη και το πόσο νερό είναι διαθέσιμο εκεί και την αναμενόμενη χρήση του ύδατος ε, για τη γεωργία, για τις μεταφορές, ε, για τις ανάγκες των πόλεων κτλ. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δούμε που υπάρχουν ανισορροπίες και τι μπορούμε να κάνουμε για να εξορροπήσουμε περισσότερο την κατάσταση. Επίσης ε, θα πρέπει να θέσουμε κάποιες ενδείξεις ε, για στόχους αποδοτικότητας ε, του νερού. Πιστεύουμε ότι οι στόχοι αποδοτικότητας για διάφορους τομείς αλλά και η βελτίωση, η βελτίωση της ποιότητας του νερού θα είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Κάτι ακόμη στο οποίο εργαζόμαστε είναι η συμπρέξη καινοτομία. Για το νερό θα συνεργαστούμε με την βιομηχανία για να αναπτύξουμε καινοτομέ λύσεις και να ξεπεράσουμε τα προβλήματα για την καινοτομία στο τομέα του νερού. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με τους συναδέλφους του ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Έρευνας για τις συμπράξεις αυτές. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσουμε μέσω δραστηριοτήτων να βελτιώσουμε τη γνώση και να ενθαρρύνουμε την καινοτομία σε ό,τι αφορά τη χρήση του νερού. Θα δούμε και το συνολικό σύστημα διαχείρισης με δύο στόχους. Καταρχήν να διασφαλίσουμε ότι είναι πλήρες το σύστημα διαχείρισής μας, ότι δεν αφήνουμε κενά. και όπου δεν έχουμε μόχλευση και όπου δεν έχουμε μηχανισμούς για να θέσουμε σε εφαρμογή τις πολιτικές μας. Αλλά παράλληλα έχουμε και την άλλη όψη του νομίσματος, η οποία είναι να μειωθεί το δικαιωτικό άχθος. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε εργαλεία πολιτικής, αλλά φυσικά θα αναζητήσουμε τα λιγότερο δαπανηρά και αυτά που επιφέρουν το μικρότερο άχθος ε, στις εταιρείες, στους χρήστες. Πρέπει να εξεύρουμε λοιπόν αυτή την ισορροπία. Έκτη προτεραιότητα. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα αυξήσουμε τη βάση, την, συγγνώμη, τη βάση δεδομένων για τις γνώσεις μας Μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους θα έχουμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε αυτά τα 170 σχέδια διαχείρισης των λεκάνων απορροής που καταθέτουν τα κράτη-μέλη τις ε, πιο σημαντικές ε, λεκάνες απορροής των ποδαμών στην Ευρώπη. αυτές οι 170 λεκάνες απορροής θα αξιολογηθούν και θα δούμε τι, ποιες τοπικές ιδέες υπάρχουν για τη χρήση του νερού σε αυτές τις ε, λεκάνες απορρίσεις των ποταμών. Και νομίζω ότι από εκεί θα προκύψουν πολλές πληροφορίες. Ε, ελπίζουμε να τις χρησιμοποιήσουμε ορθά. Πρέπει φυσικά να προβούμε και σε περαιτέρω παρατήρηση. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και το σύστημα GMES και τα δορυφορικά συστήματα για να παρακολουθήσουμε τις πιέσεις ε, στα ύδατα και να αναπτύξουμε περαιτέρω το ευρωπαϊκό σύστημα. Αυτό είναι συνεχές αίτημα από τον κύριο Ποτόστινο και τον Επιτροπό μου να διασφαλίσουμε δηλαδή ότι οτιδήποτε προτείνει η Κομισιόν βασίζεται επαρκώς σε γνώση. Οι πολιτικές δηλαδή βασίζονται σε γνώση. Σημαντικός τομέας λοιπόν αυτό. Και τέλος θα πρέπει να στραφούμε, να στραφήσουμε το βλέμμα μας και εκτός Ευρώπης πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις που θα παρουσιαστούν λόγω της λειψιδρέας ή της ε, διαθεσιμότητας του νερού, να πρέπει να δούμε την επιτεύξη των ε, στόχων της χιλιετίας και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή κατάσταση της ε, λειψιδρίας αλλά οι δημογραφικές εξελίξεις μας λένε ότι αυτά τα προβλήματα λεψιδρίας ε, θα αυξηθούν σημαντικά στο μέλλον. Αυτό είναι το σύνολο των στοιχείων ε, που θα συμπεριλάβουμε σε αυτό το σχέδιο, στο blueprint. Μέχρι την ε, εκπόνηση του σχεδίου, ε, θα έχουμε το έτος ε, του νερού και την πράσινη εβδομάδα θα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα για το νερό και την άνοιξη του 2012. Θα οργανώσουμε μια μεγάλη διάσκεψη για το είδωρ για να συζητήσουμε και όλα αυτά τα θέματα πέρα της πράσινης εβδομάδας. Πάρα πολλές ευκαιρίες λοιπόν το επόμενο έτος για να έχουμε περαιτέρω ανταλλαγές απόψεων, να καθορίσουμε καλύτερα τις πολιτικές μας. Νομίζω ότι είναι τεράστιες οι προκλήσεις, αλλά νομίζω ότι συνειδητοποιούμε όλο ένα και περισσότερο τι διακυβεύεται και έχουμε μία σειρά μέσων στα χέρια μας, τα οποία θα πρέπει να διερθωθούν με ένα συνολικό τρόπο. Σας ευχαριστώ. Äh, e Μάλιστα σας ευχαριστούμε για αυτά τα οποία μας περιγράψατε για την πολιτική του ύδατος. Η κιανοτυπία αυτή που σας αναφέρατε είναι πολύ ενδιαφέρουσα με τα διάφορα στοιχεία. Βλέπω πως απασχολείστε. Ξέρετε και η Επιτροπή μας ασχολείται πάρα πολύ εντατικά με τα ζητήματα αυτά. Το νερό είναι θεμελιώδες, ε, ουσιώδες και θα παραμείνει τέτοιο. Αναμένουμε λοιπόν την κυανοτυπία σας αυτή και έχουμε συζήτηση. Ο απόλυτος ειδικό εδώ πέρα είναι ο Ρίχαρτ Ζέμπερ και θα λάβει και τον λόγο πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, πρώτος, πρώτος ζήτησα τον λόγο. Όχι, όχι, όχι. Ε, εντάξει. Δεν θέλω... Ναι, ναι. Η Αγιάλα Σέντερ, λέει ο πρόεδρο, ζήτησε πρώτο λόγο. Ευχαριστώ να δώσω το προβάδισμα συνάδελφο. Δεν επιμένω. Ε, εν πάση περιπτώσει ευχαριστούμε τον κύριο Γενικό Διευθυντή. Χαρήκαμε για το ότι ήρθε εδώ πέρα αυτό προσώπος να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Είναι βασικό θέμα για το μέλλον και Δεν περιμένουμε ε, τις αξιολογήσεις, αλλά την και αυτή, όπως είπατε. Ο Επίτροπος ο κύριος Ποτότσνικ είχε υποσχεθεί μια σχετική ακρόαση. Εντάξει, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, αλλά ελπίζω τουλάχιστον να είναι πολύ σωστά προετοιμασμένη και από ό,τι είδα από τα διάφορα έγγραφα ε, κουράζεται πολύ η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος για να το προετοιμάσει σωστά. Μία μικρή ακόμα επιθυμία. Μέχρι στιγμής εμείς στο Κοινοβούλιο δεν ε, έχουμε εμπλακεί τόσο πολύ. Ξέρω πως έχετε προγραμματίσει διασκέψεις, αλλά ελπίζω πως ε, και νομίζω πως ειδικά το θέμα του νερού είναι τόσο ευρύ, έτσι ώστε για την κοινοτυπία αυτή καλό θα ήταν το Κοινοβούλιο να είναι στην πρώτη γραμμή. Γιατί ξέρετε υπάρχουν πολιτικές επιπτώσεις που συνδέονται και δεν είναι σε επίπεδο υπαλλήλων που μπορεί να είναι ειδικοί αλλά υπάρχουν και πολιτικά ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Οπότε ζητάω από το Γενικό Διευθυντή να εξετάσει εάν υπάρχει η δυνατότητα να μας ενημερώνει συνεχώς ως Επιτροπή. Για να συνεισφέρουμε και εμείς καμιά πολιτική ιδέα ως πρόεδρος της ομάδας Ήδατος, στην οποία είναι μέλος και η Ίνες. Θα παρακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία οπωσδήποτε και, και είμαστε στη διάθεσή σας για την περαιτέρω συζήτηση. Κάποια έτσι, βασικά ζητήματα, όπως είπατε όταν μιλάμε για νερό, ακούμε την διαχείριση της ζήτησης από πλευράς κομισιών. Θα πρέπει να δούμε αυτή την ολιστική προσέγγιση, γιατί αν συγκεντρωθούμε μόνο στη ζήτηση, δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Αν σκεφτούμε και την Κύπρο και όλο το νότιο ημισφαίριο, τα προβλήματα αυτά δεν λύνονται μόνο με τη διαχείριση ζήτησης. Ρεαλιστικά αν το δούμε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε τι άλλες λύσεις μπορούμε να έχουμε. Δεν είναι ανάγκη να έχουμε κακή θέληση των περιφερειών και των αγροτών και της κοινωνίας, αλλά θα πρέπει να κοιτάμε τα πράγματα όσο δυνατόν ευρύτερα και όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν. Όσον αφορά τώρα την περιφερειακή διάσταση, ελπίζω η Κομισιόν να τη βγάλει από την καινοτυπία που προετοιμάζει, γιατί Ίσως ε, εάν ε, δεν λάβουμε υπόψη τις τοπικές συνθήκες και γράψουμε μόνο αυτές τις φοβερές λέξεις όπως ε, διαχείριση ζήτησης, δεν, δεν θα το αντιληφθεί κανείς, ούτε πρόκειται κανείς τώρα να πάει να αγοράσει μια καινούρια κεφαλή ντους που θα είναι πιο οικονομική με το νερό για να μειώσει κατά 2% την ε, κατανάλωση. Πρέπει και εμείς λοιπόν να τα δούμε αυτά τα πράγματα ως βουλευτές αυτών περιεχών για να υπάρχει πολιτική αποδοχή αυτού του ζητήματος. Όσον αφορά την ένταξη στις λοιπές πολιτικές, κύριε Γενική Διευθυντά, γνωρίζετε ποιοι είναι αυτοί που λαμβάνουν τα πολλά λεφτά. Είναι η πολιτική, η γεωργική και ε, η πολιτική η περιφερειακή. Οπότε τώρα είναι η ευκαιρία να δούμε μέσω της διαχείρισης χρήσης γης το πώς ε, θα μπορέσουμε να καλύψουμε και τους αγρότες καθώς η γεωργία είναι ο βασικός χρήστης ε, του νερού. Ξέρω πως υπάρχει αντίσταση, είναι σαφές, αλλά το να κάνουμε μόνο ένα σχέδιο το οποίο θα βγει το 2012 και να έχουμε ήδη καθορίσει το που θα πάνε 80% των χρημάτων της Ένωσης δεν έχει πολύ νόημα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν και τα κονδύλια. Αν είναι να τα χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά πρέπει να γίνει τώρα. Και ειδικά η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και ο κύριος Ποτότσνικ θα πρέπει να μιλήσουν. Να περιμένουμε δηλαδή να ληφθούν οι αποφάσεις και να πούμε μετά mainstreaming ε, θα είναι πολύ αργά. Οπότε ξέρουμε όλοι τις εντάσεις που υπάρχουν ειδικά στον τομέα της ε, γεωργίας, οπότε πρέπει να κινηθούμε νωρίς. Όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα αρμοδιότητας και τα λοιπά, εντάξει γίνεται λόγος για περιφερειακή διάσταση και για τη χρήση γης και τα λοιπά οπωσδήποτε πρέπει να δούμε ξεκάθαρα το τι είναι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά κρατών και περιφερειών. Υποθέτω δηλαδή πως θα κατεβάσετε μια πρόταση η οποία θα είναι νομικά σωστή. Αλλιώς θα συζητάμε για αρμοδιότητα, ποιος επιτρέπει να το κάνει κτλ. Και ακριβώς στον τομέα της χωροταξίας Έχουμε μεγάλα προβλήματα και εντό των κρατών μελών. Κανία περιφέρεια δεν μας επιτρέπει να πάρουμε αυτές τις αρμοδιότητες. Οπότε θα πρέπει να διαχωρίσετε τα πράγματα από νομική σκοπιά. Αλλιώς θα μπλεχτούμε σε μία συζήτηση περί αρμοδιότητας και δεν θα γίνει τίποτα. Για την τιμή του νερού, ε, μιλάω λίγο, έχουμε λίγο χρόνο. Για την τιμή πρέπει να προσέξουμε. Το νερό, το αναφέρει και η οδηγία η σχετική, λένε πως δεν είναι απλό οικονομικό αγαθό. Και το να λέμε τώρα θα κάνουμε πολιτική με την τιμή δεν είναι σωστό. Έχουμε μιλήσει για δικαίωμα στο νερό. Αν είναι να πενταπλασιάσουμε την τιμή, Ξέρετε, θα, περιβαλλοντικά αποτελέσματα θα είναι μηδέν, θα είναι ακραία όμως τα κοινωνικά αποτελέσματα. Οπότε πρέπει να δούμε την τοπική και περιφερειακή πολιτική εδώ πέρα, γιατί, εντάξει, τιμή, ναι, ε, πολιτική τιμή, αλλά πολύ προσεκτικά με την απαραίτητη ευαισθησία. Συνολικά τώρα, ε, για την... Ε, για να βασιζόμαστε στη γνώση, συμφωνώ πράγματι έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε και εξαγωγικές επιτυχίες και μην ξεχνάμε το πρόβλημα του νερού το οποίο υπάρχει ε, ενσωματωμένο σε διάφορα προϊόντα τα οποία εισάγουμε ως Ευρωπαίοι. Πρέπει να δούμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα του ενσωματωμένου νερού σε διάφορα προϊόντα. Σημαντικό για μας και τους γεωργούς. Κάτι ακόμα αυτά, Κάτι ακόμα. Σας παρακαλώ να περάσετε στις ε, μεταρρυθμίσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να έχουμε κάτι έγκαιρα. Αν έρθει πάρα πολύ αργά δεν θα ξημεύσει κιόλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ε, συγγνώμη γιο κιόλας που ε, ή φάρμαξα την εξουσίως. Δεν πειράζει, ήταν συναρπαστικά όλα αυτά. Τα είπε ό,τι είχε να πεις, ξαλάφρωσε. Κάποιο σχόλιο εκτός μικροφώνου. Ναι, ναι, μα ξέρουμε πόσο σε απασχολεί το νερό. Πράγματι, καλό είναι κάποιος να μπορεί να, να ασχοληθεί και με αυτό το θέμα. Και οι Ινές είναι στην ομάδα αυτή ε, εργασίας. Έχει, λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή κ. Φάλκεμπερκ γιατί μας ε, συνόψε την ε, τρίτη έκθεση αλλά ταυτόχρονα εμβάθυνε σε μερικά πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. Συμφωνώ με τον κύριο Σέμπερ ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση και στην συνέχιση, στην παρακολούθηση αυτού του προγράμματος, ε, για αυτό το blueprint που περιμένουμε, το σχέδιο. Γιατί όντως είχαμε μεγάλη λειψιδρία που φάνηκε ιδιαίτερα με τις κλιματικές αλλαγές αλλά διαπιστώνουμε ότι και ο τρόπος κατανάλωσης του ύδατος δημιουργεί προβλήματα. Στην πρότασή σας λέτε να, πάρω, να λάβουμε υπόψη και άλλους τομείς πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, η γεωργική πολιτική. η γεωρική πολιτική όλο δυσάρεστες ε, ειδήσει και χαρακτηρισμούς επισύρει. Αλλά θα επικεντρωθούμε μόνο στην ε, γεωργική πολιτική. Γιατί να μιλήσουμε και για άλλες πολιτικές, όπως την ενέργεια, τη βιομηχανική πολιτική, γιατί και αυτές οι πολιτικές θα έπρεπε να αναλάβουν ένα τμήμα του βαρούς απόδειξης. Γιατί ε, για, επιρρύπτουμε όλη την ευθύνη στους γεωργούς που τους θεωρούμε ενόχους για όλα. Θα μπορούσαμε λοιπόν ε, να πούμε ότι όταν μιλούμε για εισαγωγέ, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το blueprint των εισαγόμενων προϊόντων. Για να γνωρίζουμε ποια είναι τα δεδομένα και να διευκρινίσουμε ότι μιλούμε και για άλλους τομείς πλην της γεωργίας. Μιλήσατε για εκτεταμένες διαβουλεύσεις, μιλήσατε και για διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως ξέρετε, ενδιαφέρονται όχι μόνο οι βιομηχανικοί κλάδοι, αλλά και πολλές οργανώσεις. Οργανώσεις των πολιτών, γιατί το θέμα του νερού είναι πολύ ευαίσθητο. Μας ενδιαφέρουν όλες οι καλές πρακτικές διακυβέρνηση ό,τι αφορά τις δημόσιες διαβουλεύσεις. Όλα αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν ε, στις διαβουλεύσεις ώστε όταν, όταν εμφανιστεί το σχέδιο να μην βρεθούμε προτελεσμένο γεγονότων και να μην ε, κάνουμε βεβαιασμένα τη διαβούλευση. Βέβαια, όταν ε, μιλούμε για διαβούλευση μας λένε ότι είναι χρονοβόρα διαδικασία πάντα, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν μηχανισμοί που τους έχουμε χρησιμοποιήσει σε άλλες περιπτώσεις που διευκολύνουν τη διεξαγωγή των διαβουλεύσεων. Μιλήσατε και για τις τιμές. Είπατε ότι ορισμένα από τα νέα μέτρα θα είναι και κανονιστικού χαρακτήρα. Αναφερθήκαμε στις τιμές. Υπάρχει και το θέμα το κοινωνικό που μας απασχολεί ιδιαίτερος μιλήσατε για την ε, αποδοτικότητα του ύδατος και έχουμε και ένα πειραματικό σχέδιο ώστε να ληφθεί υπόψη όχι μόνο η αποδοτικότητα των κτηρίων ως προς το νερό, πολύ αξιέπαινος ο στόχος, αλλά και η αποδοτικότητα των πόλεων ως προς το νερό. Είχαμε και στην Ισπανία κάποια στοιχεία σχετικά. Μια και λοιπόν ξεκινά και η τη συζήτηση για τις δημοσιονομικές προοπτικέ, τα διαρθρωτικά ταμεία, το Ταμείο Συνοχής, για ταμεία που επηρεάζουν πολλές πολιτικές. Πώς αυτή τη συνεκτίμηση, το mainstreaming που επισήμανε ο κύριο Σέμπερ, μπορούμε να το συμπεριλάβουμε και σε αυτά τα διαρθρωτικά ταμεία. Στην πατρίδα μου, ο εξυγχρονισμός των σωλήνων νερού εξαρτήθηκε, από τον εξυγχρονισμό των σωλήνων εξαρτήθηκε η χρηματοδότηση της επισκευή ενός κτηρίου, της ανακαίνησης ενός κτηρίου. Τέθηκε ω όρο αυτός ο εξυγχρονισμό των υδάτινων σωλήνων προκειμένου να χορηγηθεί χρηματοδότηση για μια ανακαίνιση. Θα μπορούσαμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα των δράσεων και των νέων προτάσεων για το νερό, για την για, τον, την εξασφάλιση του ανεφοδιασμού και για την εξοικονόμηση θα μπορούσαμε να τα περιλάβουμε στη στρατηγική του 2020. Και τα μέτρα που θα προτείνετε να έχουν ένα σκέλος οικονομικό, δηλαδή μείωση του σημαντικού κόστους και κυρίως ελάφρυνση του απλού πολίτη, όπως έγινε και με τον ηλεκτρισμό, με το ηλεκτρικό ρεύμα. Το ίδιο να γίνει με το νερό. Να μην πούμε ότι ε, πρέπει να εξοικονομήσετε νερό, ε, να το αναφέρουμε σε επιταγή, αλλά να, να επισημάνουμε το οικονομικό κόστος που θα έχει η μη εξοικονόμηση του νερού. Γιατί πολλές είναι, πολλά είναι τα δυσάρεστα νέα από την εξοικονόμηση, από την αύξηση των τιμών, από την αναζήτηση από τράγων ή ενόχων και στην ε, Ισπανία που έχουμε τις, ε, την αυτοδιοίκηση περιφέρειας κατηγορούμε το κεντρικό, την κεντρική διοίκηση μερικές φορές αλλά θα πρέπει να βρούμε και κάποια θετικά στοιχεία γιατί έχουμε και νέες τεχνολογίες, νέους τρόπους διακυβέρνησης που θα δημιουργήσουν και νέες θέσεις απασχόλησης πιο φιλοπεριβαλλοντικές και άρα θα οδηγήσουν οικονομική ανάπτυξη. Γιατί αν δίνουμε συνέχεια ε, κακέ ειδήσει για αυξήσει και φόρου ε, να δίνουμε και κάποιε χαρμόσυνε ειδήσει για κοινωνικά προνόμια ή κάποια κοινωνικά ενάψματα και κίνητρα. Αλλιώ, άμα μένουμε μόνο στις ε, δυσάρεστε ειδήσει, θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει αποδεκτά αυτά τα μέτρα. Ευχαριστώ. Είστε και οι δύο στην ομάδα εργασία νερού. Λοιπόν, όσοι δεν είναι τώρα στην ομάδα εργασία θα μιλήσουν λιγότερο. Γιολάντα Χιούμπνερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε το Γενικό Διευθυντή για τις, την παρουσίαση αυτής της έκθεσης για τη λειψιδρία και την ξηρασία. Σίγουρα το νερό είναι ζωτικό αγαθό και οικονομικό αγαθό και διατροφικό αγαθό για τον άνθρωπο μπορεί να είναι και πηγή ενέργειας, χρησιμοποιείται με διάφορο τρόπο και σε πολλές βιομηχανίες. Έχει πολλαπλή λοιπόν χρήση αυτό το νερό, αλλά χρησιμοποιείται και ως βασικό στοιχείο, θεμελιώδη στοιχείο της γεωργικής παραγωγής. Γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη έχει προβλήματα με το νερό, έχει λειψιδρία και ξηρασία, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε πλεονάσματα υδάτος. Και δεν έχουμε αρκετές πληροφορίε για αυτή την περιφερειακή διαφοροποίηση, γιατί προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τη λειψιδρία, αλλά με, έχουμε και τις τεράστιε τεράστιες που ήταν άνευ προηγουμένου στο παρελθόν σε ορισμένες περιοχές που ανέκαθεν είχαν πλεονάσματα ύδατος. Τώρα ακόμη και αυτές οι περιοχές αντιμετωπίζουν ξηρασίες. Μήπως θα πρέπει να επεξεργαζόμαστε κάποια στοιχεία για την αποθήκευση εμ, είδατος κατασκευάζοντας δεξαμενές για τη συλλογή είδατος. Έχουμε οδικό χάρτη ε, για τις ε, οδικές υποδομές. Έχουμε οδικό χάρτη για την ενέργεια και για τα, τους διάβλους ε, της ενέργειας. Μήπως θα έπρεπε να δημιουργήσουμε και ένα δίκτυο υδάτινο, δίκτυο με βάση τις ε, δεξαμενές, ένα οδικό χάρτη με δεξαμενές αποθήκευσης, ώστε να υπάρξει μια ισορρόπηση μεταξύ των περιοχών που έχουν πλεονάσματα και των περιοχών που έχουν λειψιδρία. Είναι δύνατο στις σύγχρονους καιρούς που έχουμε την τεχνολογία στη διάθεσή μας αυτό το θέμα να το αφήσουμε κατά μέρους, γιατί είναι προτεραιότητά μας όχι μόνο η ενέργεια, αλλά και το νερό. Θα πρέπει το στοιχείο αυτό να το εντάξουμε σε μια πανευρωπαϊκή στρατηγική για το είδωρ. Γιατί και καλύτερη διαχείριση θα κάνουμε έτσι. Θα δημιουργήσουμε και θέσεις απασχόλησης. Θα αξιοποιήσουμε καλύτερα τις διάφορες περιφέρειες που εξαιτίας της ξηρασίας της λειψιδρίας που τους μαστίζει δεν μπορούν να αξιοποιηθούν γεωργικά. Έτσι θα μπορούσαμε να αναβαθμίσουμε και αυτές τις περιοχές. Μήπως λοιπόν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πανευρωπαϊκό οδικό χάρτη να δούμε πώς έχει κατάσταση στις διάφορες περιφέρειες, γιατί πραγματικά αυτό το σημείο του νερού είναι για όλους μας ζωτικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να μην χρειάζεται κανένα αγωγός από την Πολωνία μέχρι την Πορτογαλία και να έχει αρκετό νερό η Πολωνία μέσα της καλής πολιτικής. Λοιπόν, Βιτόριο Πρόντι. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά που παρευρίσκεστε εδώ. Πιστεύω ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ε, έχουμε και την διευθύνουσα ε, ομάδα για την κλιματική αλλαγή και εγώ νομίζω ότι θα πρέπει ε, η διαχείριση του εδάφους θα πρέπει να βάλει στο επίκεντρο και το θέμα του νερού έτσι ώστε να έχουμε το νερό εκεί όπου βρίσκεται για όσο το δυνατό περισσότερο δυνατό χρόνο και για να νεώνονται τα υπόγεια ύδατα. Εγώ νομίζω ότι λοιπόν πρέπει να δώσουμε στην προτεραιότητα στο θέμα αυτό. Και θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι κυρίως στις αστικές περιοχές ε, κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο και έχουμε ε, πάρα πολλά ε, επεισόδια σε ό,τι αφορά την γιατί ξέρετε πάρα πολύ ότι επειδή μπαζώνουμε πολύ στις πόλεις δεν μπορούν να ανανεωθούν τα υπόγεια ύδατα υδροφόροι ορίζοντες και ε, δεν μπορεί το έδαφος να διατηρήσει τα ε, χαρακτηριστικά του. Έτσι λοιπόν ε, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, πρέπει πρωταρχικά πολύ δύσκολη να εξετάσουμε το θέμα της ανανέωσης των υπόγειων υδάτων και θα πρέπει επίσης ε, να έχουμε ε, μια θετική τέτοια ανανέωση, δηλαδή οι φυσικοί μηχανισμοί ίσως να μην επαρκούν. Έτσι λοιπόν ε, θα πρέπει και εμείς να παρέμβουμε σε αυτή την ενωνέωση του υδροφόρου ορίζοντα. Αυτό θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε κυρίως ό,τι αφορά τα ύδατα στις πόλεις θα έπρεπε να δούμε πώς ε, διαφοροποιούμε μεταξύ ε, των λιμάτων και ε, των όμβριων υδάτων έχουμε και και τα απόβλητα τα οποία ουσιαστικά έχουν μια περιεκτικότητα σε ενέργεια και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη βιομηχανία. Έτσι λοιπόν, αν πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ε, πρόκειται για ένα αγαθό το οποίο θα πρέπει και να παρέχεται. Το νερό θα πρέπει λοιπόν να παρέχεται. Έτσι πιστεύω ότι η στρατηγική της Κομισιόν πρέπει να εξετάσει και το θέμα της ανανέωσης των υδρόφορων ε, οριζόντων. Πρέπει να συμπεριλαμβάνεται λοιπόν τον λόγο ζήτημα γιατί νομίζω ότι πρέπει να βρούμε μια επαναξισορρόπηση μιας κατάστασης η οποία συνεχώς επιδεινώνεται. Πράγματι είναι και αυτό μεγάλο θέμα. Λοιπόν, Κρίστα Κλάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη γιατί πράγματι οι ειδικοί για το νερό τα είπαν τα θέματα να αναφερθώ εγώ σε κάτι που ενδιαφέρει εμένα. Το ότι βλέπουμε το νερό έτσι, συνολικά είναι σημαντικό για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο στο ότι είναι κάτι το σημαντικό, αλλά να ε, υπενθυμίσω ξανά την περιφερειακή προσέγγιση. Έχουμε εδώ πέρα τους συναδέλφους από τα νησιά, τη Μεγάλη Βρετανία, ας πούμε, την Ιρλανδία, δεν αντιλαμβάνονται ότι χρειάζεται κοινή στρατηγική. Πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Οι χώρες οι οποίες έχουν νερό έχουν διαφορετικά προβλήματα με τη χρήση του νερού και σε σχέση με τις χώρες που υπάρχει ξηρασία. Γι' αυτό παρακαλώ να δείτε διαφοροποιημένα αυτή τη στρατηγική και τη διαχείριση ύδατος για τις χώρες που δεν χρειάζεται να κάνουν αποταμίευση αλλά μπορούν να διαχειριστούν διαφορετικά τον Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο επίσης κύριε Πρόεδρε. Ακούστηκε πολλές φορές πως είναι καταναλωτές νερού οι γεωργοί. Κύριε Φάλγενμπεργκ, ε, παρακαλώ να αναφέρετε τους αγρότες ως τους ανθρώπους που φιλτράρουν το νερό. Πρέπει να συμπεριληφθεί αυτό στη στρατηγική του εδάφους, στη διαχείριση γης. Γιατί χωρίς το φιλτράρισμα αυτό δεν θα υπάρχει και υγιεινό νερό στα υπόγεια ύδατα για να μπορέσει ο κόσμος να στηρίξει και τους αγρότες για να συνεισφέρουν και αυτοί. Ευχαριστώ και Καλεμπάχ σαν τέλος. Μία πτυχή να τονίσω κι εγώ να συμφωνήσω με τον κύριο Πρόντι δεν είναι ανάγκη να μπούμε πράγματι στον τομέα της ε, χωροταξίας, Αλλά τι συμβαίνει, το ε, έδαφος δεν είναι διαπερατός της πόλης ε, και τι γίνεται, έχουμε κάποιες πλημμύρες που δεν θα, θα μπορούσαμε να τις έχουμε αποφύγει εάν δεν ήταν παντού το έδαφος σφραγισμένο, ναι, αν θέλετε, και ήταν έτσι κάπως πιο διαπερατό. Το έδαφος πρέπει να απορροφά το νερό, όχι να το μεταφέρουμε αλλού και να ταλαιπωρούνται περισσότερο τα οικοσυστήματα. Γιατί θα αυτοκαθαρίζεται και το νερό. Νομίζω ότι θα, το, θα τα φρόντιζε αυτά η φύση αν την αφήναμε. Μάλιστα, μία ερώτηση για το σύστημα διακυβέρνησης. Γιατί εκεί πέρα πρέπει να πούμε και εμείς κάτι για την οργάνωση του είδατο από πλευρά κομισιών. Ξέρουμε πως σε πολλέ χώρε οι κοινότητε, οι δήμοι, ε, δηλαδή είναι αρμόδιοι για αυτά, θα πρέπει να παραμείνουν ή θα πρέπει να αλλάξει αυτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αν ε, μας τα πείτε εσείς ε, σύντομα θα περάσουμε και στα, και στα υπόλοιπα. Θα προσπαθήσω. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για τις πολλές ερωτήσεις και την αντίδραση. Νομίζω λοιπόν πως συνολικά Βλέποντας ε, και αυτά τα οποία άκουσα, νομίζω πως όλοι πηγαίνουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτά τα οποία αναφέρατε περί ε, του να σκεφτούμε πέρα από τη διαχείριση της ζήτηση και για εμένα είναι σημαντικό. Πρέπει να συνεχιστεί όμως η διαχείριση της ζήτηση είναι κάτι το σημαντικό. Πρέπει πρώτα να προσπαθήσουμε να διαχειριζόμαστε λογικά το νερό πριν ε, σκεφτούμε το πώς ε, θα βρούμε περισσότερους υδάτινους πόρους. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να το δούμε συνολικά το ζήτημα, το θέμα και εμείς, οπωσδήποτε είναι σαφές πως ε, υπάρχουν μεγάλες ε, περιφερειακές διαφορές. Νομίζω τώρα αυτό με την κεφαλή του Ντούς ήταν πρωταπριλιάτικο αστείο του γερμανικού ε, τύπου και εγώ δεν μπόρεσα με στη γενική μου διεύθυνση να βρω που υποτίθεται ότι θα γίνονταν κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε συζητήσει κάτι τέτοιο. Αλλά όπως ε, ξέρετε τώρα τα μέσα γράφουν κάτι τέτοια. Δεν είναι θέμα διατάξεων και θα διατάξουμε εμείς ε, με τι θα κάνουν τους οι Ευρωπαίοι. Αλλά από κοινού μαζί με τις ε, περιφερειακές αρχές θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα διαχειριστούμε καλύτερα το νερό το οποίο είναι ένα πεπερασμένο αγαθό και νομίζω όλοι οι οι βουλευτές συμφώνησαν πως πρέπει να το διαχειριστούμε σωστά. Αλλά ταυτόχρονα να υπενθυμίσω πως παρόλες τις περιφερειακές διαφορές με το νερό έχουμε και σοβαρά διασυνοριακά προβλήματα. Και οι αρμοδιότητες, είπατε πως ε, πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και από νομική σκοπιά πάντα το κάνουμε αυτό αλλά νομίζω πως δεν θα γίνει αυτό χωρίς αντιπαράθεση αν δούμε τις δυσκολίες που υπάρχουν τώρα σε κάποια κράτη-μέλη για να κάνουν ένα σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ε, ποταμού ε, που είναι πάρα πολύ κατακαιρματισμένες οι δραστηριότητες. Εάν δούμε ταυτόχρονα π.χ. στον Δούναβο, στη, στη λεκάνη του Δούναβη που έχουμε πάρα πολλές χώρες που έπρεπε να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο γιατί μόνο από κοινού μπορούμε να διαχειριστούμε το Δούναβη ή σε πολλά άλλα ποτάμια να κάνουμε μια διαχείριση λογική και να έχουμε μια έτσι, λογική κατανομή του ύδατος για τις διάφορες ε, χρήσεις, ε, τουρισμό, γεωργία, βιομηχανία, μεταφορές, παραγωγή ενέργειας κτλ. κτλ, κτλ χρειάζεται αυτή η ευρύτερη συνεργασία και βλέπουμε ήδη με ελάχιστε εξαιρεσει και στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ανέφερα αυτό και στην ε, εισαγωγή μου υπάρχει στην ε, έκθεσή μας ε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή προβλήματα. Λειψιδρία στο Ηνωμένο Βασίλειο είπε πως υπάρχει το σοβαρότερο πρόβλημα που είχε αντιμετωπίσει ποτέ. Ταυτόχρονα και αυτό είναι το κάπως προβληματικό ζήτημα. Αν δούμε έξω από το παράθυρο πάλι βρέχει εδώ. Και το Βέλγιο ε, έχει προβλήματα λειψιδρίας. Ενώ βρέχει. ενώ αλλού υπάρχει πάρα πολύ νερό. Περνάμε λοιπόν σε μια φάση όπου η λειψιδρία ε, θα υπάρξει κατά τόπους σε ολόκληρη την Ευρώπη και ταυτόχρονα θα έχουμε πλημμύρες. Αυτό είναι και αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, ε, είναι αποτέλεσμα των ε, σοβαρών αλλαγών ε, που λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη και αλλού και εδώ πέρα νομίζω πως πρέπει να το δούμε αυτό το ζήτημα, να το καταλάβουμε καλύτερα, να καταλάβουμε τι ρόλο παίζει το έδαφος. Πρέπει να δούμε δυνατότητες ε, αποθήκευσης του νερού. Επιταχύνεται ο κύκλος του νερού που ξέρετε είναι εξάτμιση, βροχή και ξανά στη θάλασσα επιταχύνεται ο κύκλος γιατί και εμείς ε, κλείνουμε όλο και περισσότερο χώμα όπως είπατε, αποδασώνουμε και άρα έτσι η δυνατότητα συγκράτησης νερού από το, εδάφος και, από το έδαφος ε, μικραίνει. Γιατί ξέρετε πως ε, οποιοδήποτε ποτάμι θάβεται και υπογειοποιείται γίνεται μετά ε, μια περιοχή όπου τρέχει πάρα πολύ γρήγορα το ε, νερό. Δεν θα ήθελα το αναφερθώ σε όλα τα σημεία. Θα έχουμε το χρόνο όταν θα δείτε το σχέδιό μας, την κυανοτυπία αυτή. Εμείς πάντως ε, θέλουμε συνεργασία με το Κοινοβούλιο, οι ιδέες σας είναι σημαντικές για εμάς. Έχουμε κάνει κάποια τεχνική προεργασία και θα πρέπει να εργαστούμε σε πολλά τεχνικά ζητήματα οπωσδήποτε, αλλά είναι σαφές ε, πως ε, είναι πολύ πολιτικό το ζήτημα όπου χρειαζόμαστε τις ιδέες σας, την συνεργασία σας και εγώ είμαι απολύτως πεπισμένος πως το επόμενο έτος και στο δεύτερο μισό αυτού του έτους ήδη θα έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες να συνεργαστούμε και η ΜΚΟ, κοινωνία των πολιτών, θα πρέπει στην διαδικασία αυτή να εμπλακεί μου λένε πως πρέπει να σταματήσω, οπότε εάν παρέλειψα κάτι, ε, τα έχω σημειώσει όλα και θα ε, επανέλθω να είστε σίγουροι. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα δεν χάνεται όπως ξέρετε, θα επανέλθουμε σε αυτά τα ζητήματα. Οι ειδικοί του νερού οπωσδήποτε θα σας ε, ξαναπροσκαλέσουν όταν ε, εκδοθεί αυτό το η και με την πράσινη εβδομάδα και με όλα αυτά θα σας ξαναδούμε. Ευχαριστούμε που ήρθατε και καλή επιτυχία. Γεια σας. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Προσοχή εκεί. Το επόμενο θέμα που έχουμε πριν τις διακοπές γιατί είναι και επίκαιρο. Και καλωσορίζω τον κύριο Μπέκε, Γενικό Διευθυντή της, ε, του Κλίματος, που θα μας πει για τις ε, εκπομπές από εναέριες θελάσσιες μεταφορές και τυχόν ε, αντιρρήσεις που υπάρχουν. Οπότε θα μας πείτε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Κύριε Γιωστολτέικε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε εδώ και σας ευχαριστώ ναι, για την πρόσκληση, για... είδα τον τίτλο ότι αναφέρεστε και στις ενέργειες και στις θελάσσιες μεταφορές. Πάντως και στους δύο τομείς οι εκπομπές μας ανησυχούν και χρειάζεται περισσότερες δράσεις. Στο θαλάσσιο τομέα δεν υπάρχει ακόμα ρύθμιση, αλλά το 2008 είχαμε ε, κάποια ρυθμίση η Κομισιόν ε, θα αναλάμβανε, θα κατέθετε μία πρόταση αν μέχρι το τέλος του 2011 οι διεθνείς οργανισμοί και συγκεκριμένα ο Διεθνής Οργανισμός Αυτιλίας δεν παρουσιάσει κάποια δράση. Έτσι λοιπόν θέσαμε αυτή την πρόθεση για το πρόγραμμα εργασίας μας του χρόνου και η Κομισιόν θα παρουσιάσει μια πρόταση εκτός ε, και αν υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδο σε διεθνές επίπεδο. Εν τω μεταξύ συνεχίζεται η προπαρασκευαστική δουλειά. η Επίτροπος ε, Κάλλας ε, διοργανώνει ε, μία πλατφόρμα και φυσικά ε, ήταν παρόντες ε, και πρόσωποι από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Έχουμε κάποιες μελέτες οι οποίες υλοποιούνται, αλλά θέλω να τονίσω ότι η Κομισιόν δεν έχει ακόμη προσδιορίσει τη θέση της ή την προτίμησή της για το ποιο μέτρο η λύση θα προταθεί μελετούμε μια σειρά ιδεών και ξέρετε ότι τα μέτρα που βασίζονται στην αγορά, όπως ε, μια εισφορά και η συμπερίληψη του στήματος ε, εκπομπών, εκπομπών του Ευρωπαϊκού Στήματος Εμπορίας Εκπομπών, είναι δύο θέματα που μελετούμε. Όπως ε, ήδη σας είπα, σε διεθνέ επίπεδο είναι περιορισμένη η πρόοδο και στο πλαίσιο του IMO και στο πλαίσιο του ΟΗΕ δεν υπάρχουν ε, ιδιαίτερε δεσμεύσει, ούτε παρουσιάζονται μέτρα, αλλά σήμερα, καθώ μιλάμε στην ε, ε, προστασία του θελασσίου περιβάλλοντο, στον IMO, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Ναυτιλία, υπάρχει μια συνεδρίαση και θα συναντηθούν και στα τέλη τη εβδομάδα και ελπίζουμε να υπάρχει μια συμφωνία για το ευρετήριο των εκπομπών, για τον κατάλογο των εκπομπών για τα πλοία. Αυτό ελπίζουμε να αποτελέσει κάποια πρόοδο. Τώρα, αν ε, η Κομισιόν ή όταν η Κομισιόν θα παρουσιάσει την πρόταση αυτή του χρόνου, θα συνεχίσει να είναι πρόταση και ελπίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο θα συνεχίζονται και ίσως ε, να τυθεί το θέμα και πώς ε, θα έχουμε καλύτερη συνεργασία μεταξύ κομισιών και διεθνών οργανισμών. Ε, και ταυτόχρονα να συνεχίσουμε δηλαδή τις ε, συζητήσεις σε επίπεδο οργανισμών οργανισμού ναυτιλίας για να δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε και εκεί. Τώρα για την ε, σενάριες μεταφορές ε, για την αεροπλοεία. Θα ότι υπήρχαν κάποιες αναφορές, κάποια άρθρα στον τύπο, ε, υπέρ κατά της διεθνής αεροπλοείας στο σύστημα εμπορίας εκπομπών και μας εκπλήσει κάπως που υπάρχει τώρα αυτή η ένταση, γιατί ολοκληρώσαμε την νομοθεσία μας 2008 ήδη με τη συναπόφαση. Έτσι λοιπόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υιοθέτησαν μία πρόταση με συντριπτική πλειοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο και με ομοφωνία στο Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν εφαρμόζουμε τώρα την ομοθέσια και σας διαβεβαιώ ότι η εφαρμογή λαμβάνει χώρα έτσι όπως είχε σχεδιαστεί. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα ε, οι πιλότοι πρέπει ήδη να υποβαλούν εκθέσεις και να κάνουν κάποιες παρακολουθήσεις και οι εταιρείε με συγχωρείτε και όλες οι εταιρείε το πράττουν. Ε, η μεταφορά στο ιστορικό δίκαιο των κρατών μελών τελικά ολοκληρώθηκε και τα δύο ε, κράτη-μέλη, η Γερμανία και η Κύπρος που απομένουν, ε, ολοκληρώνουν τώρα τη διαδικασία και την περασμένη Παρασκευή ε, το Κοινοβούλιο στη Γερμανία ενέκρινε την ε, μεταφορά της νομοθεσίας. Τώρα στην Κομισιόν προσπαθούμε να δούμε ποια είναι τα κριτήρια αναφοράς για την ελεύθερη κατανομή. Τα κράτη-μέλη πριν από το τέλη του μήνα υποτίθεται ότι έπρεπε να στείλουν τις αιτήσει και την απαραίτητη πληροφορίε. Έγινε αυτό και τώρα η Κομισιόν, το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, θα παρουσιάσει τα benchmark. Κατόπιν ε, αυτών των κριτηρίων ε, αναφοράς ε, και πριν τα τέλη του έτους θα πούμε και στις εταιρείες, τις αεροπορικές, πώς δωρεάν, δωρεάν τέτοια δικαιώματα θα πάρουν υπήρξε και μια συζήτηση που προθήθηκε καταρχήν κυρίως ε, γιατί ενελήφθη νομική δράση από δύο αεροπορικές εταιρείες των Ηνωμένων ε, Πολιτειών και των συνδικάτων τους. Την ε, περασμένη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχαμε την πρώτη ακρόαση και ο Γενικός Εισαγγελέας ξεκαθάρισε, η Γενική Εισαγγελέας ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να παρουσιάσει την γνωμοδότησή της μέχρι τις 6 τι 6 Οκτωβρίου. Έτσι αυτό σημαίνει ότι σύμφωνα με τι συνήθειε διαδικασίε, το δικαστήριο θα ολοκληρώσει την εξέταση της υπόθεσης. Ε, ε, έξι μήνες συνήθως μετά την ακρόαση του Γενικού Εισαγγελέα, αλλά μπορεί να υπάρχει και παρέκκληση. Ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα αποφανθεί επί τη ουσία έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε την υπόθεση αυτή γιατί καθώς εμείς σεβόμαστε το κράτος δικαίου, μας εξυπηρετεί το να έχουμε σαφήνεια και σε αυτή την υπόθεση. Ταυτόχρονα έχουμε διμερείς συζητήσεις, παραδείγματος χάρη με την Αμερικανική κυβέρνηση, Είχαμε μια σημαντική συνάντηση στο Όσλο πρόσφατα. Τέθηκαν εκεί αρκετά ζητήματα από την Αμερικανική κυβέρνηση και είχαμε μια καρποφόρο συζήτηση, είχαμε και εμείς αντερωτήσεις, συζητήσαμε και με την Κίνα και με τη Ρωσία. Αλλά το δίκαιο είναι να πούμε ότι είναι αρκετά πολύπλοκες οι συζητήσεις. Πρέπει να ε, περάσουμε τα δικά μας επιχειρήματα, πρέπει να τους ε, πούμε ότι είμαστε πολύ δεσμευμένοι και ε, το αρμόδιο φορέας ο ΕΚΑΟ τελικά δεν παρουσίασε κάποια νομοθεσία που να έχει νόημα και γι' αυτό ο Ευρωπαϊκός, νομοθε... Ευρωπαϊκός Νομοθέτης αποφάσισε να προχωρήσει. Έτσι λοιπόν ε, θα συνεχίσουμε να περισπίζουμε την νομοθεσία μας. Και έτσι έχει η κατάσταση σήμερα. Έτσι λοιπόν ε, τότε θα με ρωτήσετε, τι συζητάτε λοιπόν με τις χώρες που αναφέρατε, που ανέφερα. Έχουμε το στοιχείο των ισοδύναμων μέτρων στην νομοθεσία. Τα ισοδύναμα μέτρα προβλέπονται από την νομοθεσία και θα επιτρέψουν μια εξαίρεση των εισερχόμενων πτήσεων όλων των εταιριών όταν τρίτη χώρα λαμβάνει ισοδύναμα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών. Έτσι λοιπόν αυτό τους λέμε αν μια χώρα λάβει ισοδύναμα μέτρα, τότε θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε, να σκεφτούμε, να άρουμε τις υποχρεώσεις για τις ερχόμενες πτήσεις. Και σε σχέση με τον αντίκτυπο της αεροπορίας ε, πέραν του διοξιδίου του άνθρακα. Όταν λάβαμε την ε, απόφαση να συμπεριλάβουμε την διεθνή πλοία το 2008, η Κομισιόν έκανε μια δέσμευση να παρουσιάσει μια πρόταση για τους αντικτύπους πέρα από το διοξείδιο του άνθρακα και έχουμε, ξέρετε, και άλλες ουσίες όπως οξύδιο του αζότου, του θείου κτλ. Και το μελετάμε όλα αυτά. Και είναι πιο δύσκολο να προσδιορίσουμε το μέγεθος του αντικτύπου. Λαμβάνει χώρα και άλλη έρευνα στο πλαίσιο της IPCC, συγκεκριμένα. Εκεί μελετάμε και παρακολουθούμε ε, ε, εκ του σύνεγγυ τα αποτελέσματα της ε, επικαιροποίηση, αλλά είμαστε σόφρονες και θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας όταν έχουμε μία πιο σαφή εικόνα σε σχέση με το μέγεθος του δικτύπου της αεροπλοείας πέρα από το διοξείδιο του άνθρακα για τις υπόλοιπες ουσίες. Ελπίζω να κάλυψα τα περισσότερα από τα σημεία, αλλά φυσικά αν έχετε ερωτήσεις ευχαρίστω να απαντήσω. Σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Τελβέκε. Ήταν σαφέστατες οι πληροφορίες που μας δώσατε. βρισκόμαστε στο 2011 και λίγο πριν τη θέση εφαρμογή του συστήματος ε, ήδη γίνονται κάποιες απόπειρες για τορπίληση του συστήματος. Τώρα, έξι μήνες μετά την παρουσίαση των συμπερασμάτων ε, της Γενικού Εισαγγελέας, δεν ξέρω ε, τι θα γίνει. Η ΕΠΑ πάντως και η Κίνα, οι δύο μεγάλες χώρες έχουν επέμβει, αλλά υπάρχουν και πολλές μικρές χώρες Ελπίζω να μην γίνει διαφορά μεταξύ των μεγάλων και των μικρών χωρών και να μην επωφεληθούν οι μεγαλύτερες χώρες ε, εις βάρος των μικρών. Δηλαδή ε, να ωφεληθούν από το σύστημα οι μεγάλες και οι μικρές ε, να πορευθούν εκ των ενόντων. Ο Πέτερ Λίζε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση και σας ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί η απόφαση για τη θέσπιση αυτής της νομοθεσίας έγινε μετά από διεξοδική αξιολόγηση των επιπτώσεων. Και το επιχείρημα που μπορούμε να προτάξουμε είναι αντιενός ισχύει. Μόνο αν παραμείνουμε ενωμένοι θα μπορέσουμε να προσπίσουμε τα συμφέροντά μας απέναντι στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί αν σκύψουμε το κεφάλι ε, και υποχωρήσουμε μόνο και μόνο επειδή μας απειλεί η Κίνα, Νομίζω ότι δεν είναι σωστή αυτή η μέθοδος. Δεν θα πρέπει εμείς κάθε φορά που διαμαρτύρονται οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι, εμείς να αλλάζουμε την νομοθεσία. Μόνο και μόνο επειδή διαμαρτύρονται έντονα. Στις ε, Ηνωμένε Πολιτείε έχουμε 60 δολάρια φόρο που πληρώνουμε στο εισιτήριο για τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Βλέπουμε το ύψος των αεροπορικών εισιτήριων στην ε, Γερμανία, Γαλλία ή τη Μεγάλη Βρετανία. Ποια είναι τώρα τα ισοδύναμα μέτρα. Υπάρχει ήδη ένας κατάλογος για να δημιουργηθεί ένας τρόπος αναγνώρισης των ισοδύναμων μέτρων. Σε ό,τι αφορά τις αζωτούχες ε, ενώσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πολύ πιο ακριβής και υπάρχει συγκεκριμένη συμφωνία με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις μεταφορές, στο Κανκούν διαπιστώσαμε ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν από μόνο τους να σημειώσουν πρόοδο. Γι' αυτό και περιμέναμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Ζιλ Παρνιά, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γενική Διευθυντά, το σχέδιο που μας παρουσιάσετε είναι φλέγον και από οικονομική άποψη. Πριν από λίγο ακούσαμε διάφορες ε, φημολογίες, μετά μας ενημερώσατε για τις συζητήσεις που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ε, είτε για τις διαπραγματεύσει που έχουμε με τη Ρωσία και την Κίνα. Όλοι φαίνεται ότι ανησυχούν και οι αεροπορικές εταιρείε, οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείε που έχουν πληγεί από την άνευ χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Κάθε τρεις και λίγο γίνονται συγχωνεύσεις εταιρεών και οι κατασκευαστές ανησυχούν τα μάλα, γιατί η Κίνα μας λέει σήμερα ότι αν δεν αλλάξουμε το σύστημα δεν θα αγοράσουν τα Airbus μας οι Κινέζοι, αυτή είναι η απειλή τους και τα αεροδρόμια επίσης ανησυχούν γιατί ήδη γνωρίζουμε ότι κάποιες χώρες και με μερικές μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ε, δήλωσαν, ανήγγυλαν ότι θα παρακάμπτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους ευρωπαϊκούς αερολιμένες προκειμένου να ε, φτάνουν στις Ηνωμένε Πολιτείες και προτιμούν να περνάνε από τις χώρες του κόλπου. Πέραν της ε, εύλογης μας ανησυχίας για την νομοθετική δράση, η γερμανική και η γαλλική κυβέρνηση συνυπέγραψαν ε, μία επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Αρμόδιο Επίτροπο, όπου εξέταταν τις ε, σοβαρές τους ανησυχίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να μας καθησυχάσει, είπε ας μην πανικοβαλόμαστε, θα εξετάσουμε κάποια μέτρα όπως αυτά που μας παρουσιάσατε σήμερα στην ομιλία σας και γνωρίζουμε ότι, ότι και οι ενώσεις κατασκευαστών αεροπορικών εταιριών ε, έχουν προτείνει πέραν των στόχων αυτών και κάποια μέτρα. Εσείς έχετε καταρτήσει μελέτες αξιολογώντας τα μέτρα που προτείνει ο κλάδος. Ευχαριστώ. Λέω κύριο Σάικουτ. Σας ευχαριστούμε που μας δώσετε αυτή την επισκόπηση για το σημερινό για την ε, θάλασσες και ενέργειες μεταφορές, για τις ενέργειε μεταφορές. Θέλω να συγχαρώ την Κομισιόν ε, που έχουν ε, κάθε τη θέση και πραγματικά επιμένετε στην νομοθεσία επί της οποίας έχουμε συμφωνήσει. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε να καταλήξουμε κάπου. Στην αρχή όλοι είναι κάπως ε, ε, πιο αγχωμένοι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να επιμένουμε εδώ αλλά όπως είπε και ο κύριος Λίζε, τι ακριβώς εννοείτε όταν λέτε συζητάτε ισοδύναμα μέτρα, συζητάτε για ισοδύναμα μέτρα με τις μεγάλες χώρες, ε, θα μπορούσε να υπάρχει κάποια διέξοδο γι' αυτό. Αλλά από ό,τι ξέρω, εγώ ποτέ δεν έχω ακούσει για τέτοια ισοδύναμα μέτρα να λαμβάνονται στις ΥΠΕ στην Κίνα. Μήπως ε, μπορείτε να αναφερθείτε περαιτέρω σε αυτό το θέμα τώρα σε ό,τι αφορά το οξύδιο του ζώτου ε, στην νομοθεσία με σαφήνεια λέγεται ότι η Κομισιόν ήδη από το 2008 θα παρουσίαζε μια πρόταση για να καταπολεμήσει τον αντίκτυπο των οξυδίων του αζότου. Τώρα λέγοντας ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ενώμη στην έπιση, νομίζω ότι είχαμε προσχεθεί να κάνουμε κάτι στην νομοθεσία. Αναμένω λοιπόν από την Κομισιόν κάποιο πιο τολμηρή στάση εκεί. Τώρα για τις θαλάσσιες μεταφορές. Είναι σαφές ότι πιθαν, πιθανότατα χρειαζόμαστε μια πρόταση αν ή όταν θα έλθει του χρόνου και αναρωτιέμαι και για τη νομική βάση της εισφοράς. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς να το πράξουμε, είπατε, αλλά αμφιβάλλω αν αρκεί η νομική βάση για μια εισφορά και θεωρώ ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε περισσότερο τους κανόνες αγοράς γιατί για την εισφορά αν ε, μπορεί να τεθεί η βέτα από τα κράτη-μέλη θα έχουμε πρόβλημα να διορθωθεί εκεί η βάση δεδομένων και να μας πείτε τι κάνετε και με τα εισοδήματα. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, Γιος, και ευχαριστούμε για τις εξηγήσεις είναι σημαντικές. Γιατί διακούμε διάφορα στον τύπο. Να ρωτήσω κάτι. Είπατε. Ξέρετε πως ε, το επόμενο έτος ε, διάφορες επιτροπές θα ασχοληθούν με την αναθεώρηση της οδηγίας περί φορολογίας της ενέργειας. Και οπωσδήποτε κοιτάμε το θέμα του κλίματος με ενδιαφέρον. Έχετε κάποια πρόταση για τον εισηγητή της γνωμοδότησης αυτής της Επιτροπής. Έχετε κάποια πρόταση για το θέμα της ε, ναυτιλίας ε, και της αεροπορίας, για κάποιον άλλο τρόπο προσέγγισης ε, για να αντιμετωπίσουμε την άσχημη εξέλιξη σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ. Βιτόριο Πρόντι. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ τον ε, κύριο Διευθυντά. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά για την παρουσίασή σας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα φόρο που να επιβάλλεται στα καύσιμα που χρησιμοποιούν οι αεροπορικές εταιρείε. Έτσι λοιπόν ε, μέλλον έχουν κακομάθει και θα πρέπει να σκεφτούμε και μια τέτοια περίπτωση, την έλευση ενσέτειου τέτοιου φόρου. Εγώ νομίζω ότι ένα ισοδύναμο μέτρο θα μπορούσε να είναι στην περίπτωση των ΕΠΑ ένα νομοσχέδιο, το χάρη για το cap and dividend όπου αποφασίζεται ότι ουσιαστικά υπάρχει κάτι αντίστοιχο με αυτό που προτείνεται από την Ένωση, όμως στη συνέχεια τα έσοδα από εκεί ξαναδίνονται στον Αμερικανικό λαό. Από τη σκοπιά του κόστους ε, του αεροπορικού εισιτηρίου νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι κάτι ισοδύναμο. Δηλαδή να υπάρχει μια εσωτερική ανακατανομή και αυτό θα μπορούσε να ίσως και ενδιαφέρον να το διερευνήσουμε. Τώρα, πλην του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να δούμε τον αντίκτυπο αυτό, αλλά εμείς ως Ευρώπη έχουμε κάνει βήματα προς τα μπρος με τον Ευρωπαϊκό Ουρανό και τον Καθαρό Ουρανό και με τη βελτίωση των επιδόσεων των κινητήρων. Επομένως έχουμε μικρότερη εκπομπή σε οξύδιο του αζότου. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το εξής, ε, το ότι η αεροπλοεία ε, εκπέμπει στη στρατόσφαιρα ε, αυτά τα μόρια τα οποία λέγονται break carbon και αυτό μπορεί να έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό αντίκτυπο. Δηλαδή, σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στην ατμοσφαιρική στροποσφαίρα, στη στρατόσφαιρα, η περίοδος παραμονής αυτών των σωματιδίων θα μπορούσε να φτάνει και τον ένα χρόνο. Αυτό να το έχετε κατά νου. Σας ευχαριστώ. Κράτσε, Ματίας. Ευχαριστούμε. Ματίας, ναι. Ευχαριστώ πολύ για αυτά που μας είπατε κύριε Ντελμπέκε. Εμείς είχαμε συμφωνήσει τότε εγώ ήμουν σκιώδη συγητή. είχαμε συμφωνήσει με το φάκελο τότε γιατί είχαμε δήλωση της Κομισιόν πως θα έχουμε νομοθετική πρόταση για τα οξύδια του αζότου και δεν έχουμε ακόμα τίποτα. Οπότε, παρακαλώ, να υποβληθεί. Είπατε τους λόγους για τους οποίους δεν γίνεται, αλλά ούτως ή άλλως εμείς και εγώ σας υποστηρίζουμε πλήρως στον αγώνα που πρέπει να δοθεί. Και έχουμε και μεγάλη πλειοψηφία εδώ και είχαμε και στο Κοινοβούλιο για την συμπερίληψη της αεροπορίας. Το είχαμε ζητήσει. Αλλά οι τάσεις στα κράτη-μέλη, βλέπουμε εδώ και εκεί υπάρχουν διάφοροι αεροπορικοί φόροι, π.χ. είπαμε από 5,7 τόνους και πάνω. Μα, στη Γερμανία είναι και κάτι μικρά αεροπλανάκια που πάνε σε κάτι νησιά, με ένα φόρο που είναι όσο ολόκληρο το ειστήριο. Οπότε ε, έχουμε αναπτύξει ένα μέσο το οποίο ε, δεν είναι γραφειοκρατικό αλλά δεν επαρκεί και το μέσο αυτό το οποίο ε, αποφασίσαμε θα το υπερασπίσουμε με ό,τι έχουμε στην διάθεσή μας και θα σας στηρίξουμε και έτσι θα έχουμε και αξιοπιστία. Από εκεί θα εξαρτηθεί η αξιοπιστία της κλιματικής πολιτικής της Ευρώπης. Εάν υπερασπιστούμε με ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας αυτό το πράγμα. Γιατί, το είπε και ο κύριος Λίζε, τότε θα είμαστε διεθνώς αξιόπιστοι. Αλλιώς όχι. Ευχαριστώ. Τελευταίος ο Ρίχαρτ Ζεμπερ. Ευχαριστώ. Και εγώ να σας ενισχύσω κύριε Ντελμπέκε. Ειδικά πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει αποδοχή εντός της Ευρώπης και άρα δίκαιη κατανομή γιατί ξέρετε είπατε και εσείς πως αναπτύσσεται η αεροπορία και δεν πρέπει να την επιβαρύνουμε και άρα θα πρέπει οι φόροι αυτοί το επιπρόσθετο κόστος να αποδοθούν ούτως ή άλλως κάπου γιατί τα κράτη-μέλη τι κάνουν πρώτον διπλασιάζουν τους φόρους και δεύτερον δεν πάνε μετά στην αεροπορία αλλά τους παίρνουν και τους κάνουν ό,τι θένε. Οπότε νομίζω καλό θα είναι να δούμε πού πηγαίνουν μετά αυτά τα χρήματα για να ξέρει σε τι συνεισφέρει και ο, ο επιβάτης. Για τα πλοία, για την αυτιλία. Εντάξει, μπορείτε εκεί πέρα νομίζω να κινηθείτε, αλλά μην ανησυχείτε. Το να συμβεί κάτι σε διεθνέ επίπεδο πριν από το ευρωπαϊκό είναι πάρα πολύ απίθανο. Θα πρέπει όμως άρα να το δείτε πολύ προσεκτικά, ήρεμα, για να έχετε σωστή νομική βάση. Οπότε να δείτε ε, όλα τα αποτελέσματα τα οποία έχει αεροπορία, ακόμα και τα λεγόμενα θετικά στο κλίμα μέσω της αντανάκλασης λοιπά Γιατί να μην ανοίξει κανένα παραθυράκι. Βεβαίως, λέει ο πρόεδρος, ε, Δεν ξέρω πώς έχουμε καταλήξει αεροπορικές εταιρείε από άλλες χώρες να καταργούν την ομοθεσία μας και να προσπαθούν να την ε, νερώσουν. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά μάλλον θα βρεθούν κάποια στιγμή ενώπιον του ΔΕΚ στο Λουξεμβούργο. Παρακαλώ λοιπόν έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ για την υποστήριξη και εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η νομοθεσία πέρασε από πλήρη διαδικασία συναπόφασης και γι' αυτό θα πρέπει να την υποστηρίξουμε, να εμείνουμε. Το θέμα των αντιπίνων ε, και οι παραγγελίες των Airbus αναφέρθηκα στη συζήτηση. Η Airbus ε, είχε στο Λεμπουζέ μια επιτυχή εκδήλωση και δεν αναφέρθηκε σε επίσημες ε, ε, συνεδριάσει, αλλά παρασκηνιακά ακούστηκε και κάποιε φημολογίε. Α τι αφήσουμε λοιπόν σε αυτό το επίπεδο αυτές τις ειδήσει των φημολογιών, γιατί η μόνη αξία που βλέπουμε είναι το κατά πόσο η έρμπα θα κατασκευάζει σωστά αεροπλάνα ε, αποδοτικά από άποψη ε, ενέργειας και πώς θα τα θέσει σε εμπορία, αυτό που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει. Τώρα το μείζον ζήτημα στα ισοδύναμα μέτρα αφορά την αρχή που θα υποστηρίξουμε στο μέλλον στις κλιματικές διαπραγματεύσεις και είναι κάπως ατυχές ότι στην περίπτωση αυτή δεν μας υποστηρίζουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Γιατί έχουμε με βάση την, ε, τον ΟΗΕ την κοινή αλλά διαφοροποιημένη αρχή. Εδώ έχουμε έναν ε, ολοκληρωμένο κανόνα και δεν είναι μονομένες χώρες ε, που θα πρέπει να υποβάλουν τα μέτρα τους γιατί Μιλάμε για τη μέση τάξη για τους επιχειρηματίες. Έχουμε πραγματικά σφαιρικό ανταγωνισμό και η κοινή αλλά διαφοροποιημένη αρχή θα πρέπει να αποκτήσει την δέουσα αξία. Θέλουμε λοιπόν θεμητό και σταθερό ανταγωνισμό για την αγορά αυτή. Είναι σημαντικό και για την διεθνή ε, ε, το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας που θα πρέπει να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο γιατί δεν υπάρχει ρύθμιση γενικά στην αεροπορία. Ε, ιδιαίτερα σε περίπτωση που δεν πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για που δεν παίρνουν από την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τώρα την εκτίμηση των ισοδύναμων μέτρων, ο ισότιμο ανταγωνισμό μεταξύ των αεροπορικών εταιριών μα ενδιαφέρει. Και θεμητό ανταγωνισμό, ίσω ανταγωνισμό ε, και αναγνώριση ισοδύναμων μέτρων δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μια κατάσταση που θα παγιώσει προνομιακή μεταχείριση της μίας ή της άλλης αεροπορικής εταιρείας ανάλογα με τη χώρα προέλευσης της. Θα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε τα ισοδύναμα μέτρα βέβαια, την ισοδυναμία, αλλά σε άλλες περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέδειξε ότι μπορεί να προχωρήσει και στο θέμα αυτό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν υποβληθεί προτάσεις ισοδύναμων μέτρων για εξέταση. Αναφέρεται ο στόχος του 22%, περιορισμός ε, του 22% σε σχέση με τη μέχρι τώρα κατάσταση στην Κίνα. Άλλη πρόταση παρόμοια αναφέρθηκε για τις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά ανεπίσημα, δεν έχουν ε, υποβληθεί επίσημα από τις ενδιαφερόμενες χώρες και από τη στιγμή που δεν κατατεθούν επίσημα οι προτάσεις δύναμων μέτρων δεν μπορούμε και να τις αξιολογήσουμε. Ένα άλλο σχόλιο αφορά το, την οδηγία για την ε, φορολογία ενέργειας, τον ενεργειακό φόρο. Ένα σημαντικό θέμα είναι αυτό της ενεργειακής φορολογίας που δεν είναι και πολύ ελκυστικός μηχανισμός και θα πρέπει να περάσει με ομοφωνία στο Συμβούλιο. Εξού και η δυσκολία γιατί δεν υπάρχει συμφωνία. Γι' αυτό και στο παρελθόν προτιμήσαμε το, το σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου γιατί για την έγκριση τέτοιου νομοθετήματος αρκούσε η ενισχυμένη πλειοψηφία. Και υπάρχει τεράστια διαφορά στο Συμβούλιο να συνεχίζαμε στη δεκαετία του 90 τότε τη συζήτηση για το ενεργειακό φόρο του άνθρακα. Αν μέναμε στη συζήτηση αυτή, δεν θα είχαμε σημειώσει καμία περίπτωση πρόοδο. Ευτυχώ που περάσαμε στη συζήτηση για το σύστημα εμπορία εκπομπών, που διευκόλυνε πολύ την κατάσταση και πέρασε και το σχέδιο. Σε ό,τι αφορά τις εκπομπές εκτός του διοξιδίου του άνθρακα, τα σχόλιά σας θα τα μεταφέρω και στους συναδέλφους και θα τα συζητήσουμε. Πάντως το πιο σημαντικό είναι να θέσουμε ως προτεραιότητά μας να λειτουργήσει το σύστημα σε διεθνές επίπεδο. Και απομυζεί τους πόρους μας ε, περισσότερο από ό,τι περιμέναμε, γιατί έχουμε πολλά, πολλά ζητήματα, πολλές διμερείς ε, δραστηριότητες. Πάντως, ε, ως προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή και εκεί είναι που δρομολογούμε τους πόρους μας. Είναι στο σημείο αυτό. Πάντως σημείωσε και τα υπόλοιπα σχόλια της συζήτησης. Θα τα μεταφέρω στους αρμοδίους. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντελμπέκε για την παρουσίαση της έκθεσής σας. Ε, εμείς, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, είμαστε πολύ αυστηροί και δεν θέλουμε να ενδώσουμε σε σχέση με αυτά που είχαμε αποφασίσει στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, καλή επιτυχία σας εύχομαι και ραντεβού το απόγευμα. Μην ξεχνάτε ότι θα μας επισκεφθεί η Υπουργός Υγείας της Πολωνίας.